Bonjour à tous. Good morning everybody. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε. Στην ε, ακρόαση για την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χαρά μας να ε, σας ε, καλωσορίζουμε εδώ σήμερα, όχι μόνο τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και όλους τους παρισταμένους που εκπροσωπούν οργανώσεις και θεσμικά όργανα και όργανα που είναι αφιερωμένα στην αρχή της ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω αυτήν την ακρόαση, διότι είναι πάρα πολύ σημαντική λόγω του θέματός της. Αναφερόμαστε στην Ιθαγένεια, στη βασική ιδέα της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε επικεντρωθεί τόσο πολύ στις συνέπειες της κρίσης ε, που ζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάπως, κατά κάποιο τρόπο, ε, κάποιοι έχουν ε, πάψει να αντιλαμβάνονται ότι το ευρώ δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καν η ενιαία αγορά δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και αξίες της είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι αυτό το οποίο υπογραμμίζονται εδώ και 20 χρόνια, από τότε που προέκυψε η έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας στη συνθήκη του Μάστρεχτ το 1992 και μαζί της είχε και μια σειρά από συγκεκριμένα δικαιώματα που για πρώτη φορά αποτυπώνουν την ιδέα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, Να μπορεί κάποιος να μετακινείται ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην υπάρχουν διακρίσεις για λόγους εθνικότητας, κάτι το οποίο ήταν ανέκαθεν βασική αρχή της ευρωπαϊκής διαδικασίας, να μπορεί κάποιος να ψηφίζει και να είναι υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές αν και ανεξάρτητα από το που κατοικεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει δικαίωμα συνδρομής και προσφυγής σε ε, πρεσβεία ή προξενείο άλλης χώρας μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν δεν εκπροσωπείται η χώρα του. Ε, γνωρίζουμε τα προβλήματα αυτά καθημερινά, τα βλέπουμε στην Επιτροπή Αναφορών. Μπορεί κάποιος να κάνει αναφορά στον ε, Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και μπορεί να ζητήσει να οργανωθούν και να στηριχθούν ε, πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να προτείνει νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, μπορεί πλέον να απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα τα οποία αναφέρονται στη Χάρτα των ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται λοιπόν για το πιο σημαντικό ζήτημα, το οποίο εφαρμόζεται σε αυτή την εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, συμπίπτει με την έναρξη ισχύω τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Υπάρχουν μια σειρά από μέτρα τα οποία συζητήθηκαν στι διάφορε επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, οι δέσμοι μέτρων Σέγγεν, ε, τα θέματα ποινική δικαιοσύνη, δικαστική συνεργασία. Τα δικαιώματα λοιπόν που περιλαμβάνονται σε όλη αυτή τη διαδικασία, ε, η ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ενημέρωση ή ε, νομική συνδρομή. πριν υπάρξει οποιαδήποτε νομική δίωξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει το θέμα των δικαιωμάτων των θυμάτων ε, και προστασία των θυμάτων τρομοκρατίας, η ε, λεγόμενοι δέσμη μέτρων για τα θύματα. Υπάρχουν επίσης και οι διάφορες ε, προκλήσεις που αφορούν την ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυδαιμονίας παιδιών, θέματα δικαστικής συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους. Αυτό είναι βασικό ζήτημα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια υπάρχει και έχει μεγάλη σημασία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συζητάτε ιδιαίτερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παλιά έλεγα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πιο σημαντικό κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή, η συγκεκριμένη θητεία στην Ευρωπαϊκή Ιστορία. Πολλό δε μάλλον είναι το πιο σημαντικό κοινοβούλιο σε όλη την Ευρώπη. Αν το γνώριζε αυτό ο κόσμος, αν γνώριζε ο κόσμος ότι εμείς εδώ τους εκπροσωπούμε, εκπροσωπούμε 500 εκατομμύρια ανθρώπους και θα πρέπει λοιπόν να τους προσεγγίσουμε, θα πρέπει όχι μόνο να τους ε, γνωστοποιήσουμε ότι έχει σημασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά να ε, γνωρίζουν και ότι το, οι ευρωεκλογές ε, του 2014 έχουν μεγάλη σημασία η ισχύ του Κοινοβουλίου πρέπει να ενισχυθεί και ο κόσμος θα πρέπει ε, να έχει κίνητρο για να συμμετέχει και να δεσμεύεται στην ευρωπαϊκή διαδικασία. Ε, το δικαίωμα ψήφου στις εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές θα πρέπει να επισημαίνεται και να τονίζεται πόσο σημαντικό είναι και ε, να δείξουμε ότι είναι στοιχείο, αναπόσπαστο στοιχείο της ευρωπαϊκής ταυτότητας των πολιτών. Διότι μόνο έτσι θα επιτύχουμε ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όταν οι πολίτες γνωρίζουν και είναι περήφανοι για την ευρωπαϊκή τους ηθαγένεια. Ε, και η οποία συμπληρώνει την εθνική τους ταυτότητα, τα δικαιώματα που απολαμβάνουν ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο ε, και να υπάρχει ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, ώστε το θέμα της ευρωπαϊκής ηθαγένειας να είναι πλήρες. Και αυτό είναι αυτό το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα σε αυτή την ακρόση. Και σας καλωσορίζω και πάλι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και ευχαριστούμε φυσικά και την, το συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι η κυρία Φρανσουάς Λεπάη, η διευθύντρια εδώ, ε, η κυρία Ρέγνερ, η οποία εκπροσωπεί την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, η οποία ασχολείται ιδιαίτερα με τα θέματα αυτά από την νομική του σκοπιά και ε, τα θέματα αυτά συμπληρώνουν την ε, εικόνα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι υπάρχει διερμηνία σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάποιες εξαιρέσεις. Δυστυχώς δεν υπάρχουν εσθονικά, ε, φιλανδικά και μαλτέζικα. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες διατίθενται, υπάρχει διερμηνία σε όλες τις γλώσσες. Επίσης, να σας πω ότι η ακρόαση αναμεταδίδεται και καταγράφονται, μαγνητοσκοπούνται οι παρεμβάσεις των συμμετοχόντων και των ομιλητών. Σήμερα το πρωί θα επικεντρωθούμε στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας και στην ε, θεμελίωση της πολιτικής συμμετοχής ε, των Ευρωπαίων πολιτών. Το λόγο θα λάβει η συνάδελφος, η κυρία Ρέγνερ, η οποία είναι η πρώτη αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Και στη συνέχεια, ακριβώς, ε, έχουμε το πρώτο πάνελ ομιλητών και την πρώτη παρέμβαση θα κάνει η κυρία Φρανσουάζ Λεμπάιλ εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Ρέγνερ, έχετε το λόγο. Σας εύχομαι ένα πάρα πολύ καλό και ευχάριστο πρωινό. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μας, στο σπίτι σας. Είσαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είσαστε ε, στο σπίτι σας. Εγώ είμαι Αυστριακή, είμαι από, από τη Βιέννη, αλλά είμαι κυρίως ε, πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, γι' αυτό θα συζητήσουμε σήμερα ακριβώς όλα τα δικαιώματα τα οποία έχουμε λόγω αυτής της ηθαγένειας, λόγω αυτής της ιδιότητας. Έχουμε τη δυνατότητα να κυκλοφορούμε, να ταξιδεύουμε, να εργαζόμαστε χωρίς καμία διάκριση σε άλλες χώρες της Ένωσης και γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό, σημαντική η παρουσία σας σήμερα εδώ είναι βεβαίως βασικές αρχές τις οποίες πρέπει εμείς να βιώσουμε, να ζήσουμε. Και γι' αυτό εκτός από την, ε, τις ευρωπαϊκές, τα ευρωπαϊκά όργανα και οργανισμούς, εσείς είσαστε εκείνοι οι οποίοι θα μας πούνε, εκτός από την ε, Εκτελεστική Επιτροπή, την Κομισιόν, ε, τι δεν πάει καλά, τι παράπονα έχετε, τι μπορούμε να διορθώσουμε και τι άλλο πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας ως υπήκοοι ως ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να αναφερθώ στην ε, πρωτοβουλία ε, στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, η οποία δημιουργήθηκε με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Υπάρχουν βεβαίως ακόμα τεχνικές δυσκολίες στην πλήρη υλοποίηση, υπάρχουν και δημοσιονομικά προσκόμματα, αλλά η πρωτοβουλία αυτή δείχνει έντονα ε, ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να την ε, εφαρμόσουν, θέλουν να την ε, βελτιώσουν και θέλουν να βοηθήσουν σε πολλά προβλήματα τα οποία θίγουν τους Ευρωπαίους πολίτες όπως παραδείγματος χάρη πρωτοβουλίες για την παροχή κονδυλίων για την βελτίωση υποδομών. Ε, τώρα η πρωτοβουλία αυτή από ένα εκατομμύριο θα αυξηθεί ε, στα δύο εκατομμύρια ε, κατόπιν πίεσης υλοποίησης πολλών προγραμμάτων. Αυτό δείχνει ακριβώς πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις δυνατότητες της Ένωσης. Επίση, η Νομική Επιτροπή ασχολείται με προγράμματα τα οποία αφορούν ε, τις κατασκευές, τις θέσεις εργασίας στον τομέα των κατασκευών, η Επιτροπή Περιβάλλοντος με το θέμα παροχής καθαρού νερού και όλες μας ε, οι επιτροπές και ιδίως η Νομική Επιτροπή ασχολείται με νομικά δικαιώματα και την κατοχήρηση των νομικών δικαιωμάτων βάσει γνωμοδοτήσεων τη νομική υπηρεσία, διότι... Η όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή ηθαγένεια σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες μας πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, τα νομικά τους δικαιώματα και να μπορούν να τα προασπίσουν και να τα... Ε, σε περίπτωση δηλαδή που χρειάζεται δικαστική προσφυγή και να μπορούν να ξέρουν πότε πρέπει να καταγγείλουν κάποια παράβαση. Γι' αυτό ακριβώς Θέλω να αναφέρω τώρα σε έναν άλλον τομέα, στον εκπαιδευτικό, το πρόγραμμα Erasmus, Erasmus το οποίο είναι εξαιρετικά επιτυχημένο, ιδίω για μαθητευόμενους. Έχει ε, καλύψει και ο στόχος του είναι να καλύψει το μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών, μαθητευόμενων και ασκούμενων διασυνοριακά, έτσι ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εκπαιδευτικές δυνατότητες. Ο Λόπες Αγγιλάρ που είναι πρόεδρος Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών το ανέφερε ήδη. Αυτό που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι η πρόσβαση στην πληροφόρηση. Τι γίνεται στην Ευρώπη, πώς μπορούμε να πληροφορήσουμε τον κάθε πολίτη τι σημαίνει ακριβώς αυτή η ιδιότητα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Είναι ένα τεράστιο θετικό, μια τεράστια θετική ιδιότητα αυτή και γι' αυτό ακριβώς ε, θέλουμε να ακούσουμε τη δική σας κριτική, τα δικά σας σχόλια και παρατηρήσεις και θα θέλαμε να αναφερθείτε σε συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία θα σημειώσουμε και θα κοιτάξουμε να προωθήσουμε στην ατζέντα μας και γι' αυτό προσβλέπουμε μεγάλη ικανοποίηση σε αυτή την ακρόση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ρέγνερ και τώρα θα δώσω το λόγο, λέει ο πρόεδρος, στην κυρία Λεμπάη, η οποία είναι Γενική Διευθύντρια της Γενική Διεύθυνσης Δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια Πρόκειται για μια κοινή συνεργασία μεταξύ τριών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι το πρέπον είναι να προσπαθήσουμε να δούμε τι θα ήθελαν ε, οι πολίτες να συμβεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, στην Ευρώπη πριν από τις ευρωεκλογέ. Γνωρίζετε ότι το 2010 ξεκίνησε μια έκθεση για την ηθαγένεια και προτείναμε τότε 25 μέτρα για τη βελτίωση της ηθαγένειας ε, στην Ευρώπη. Στο μεταξύ έγιναν αρκετά προκειμένου να επιτευχθούν ε, όλα όσα προτάθηκαν τότε είτε για θέματα διασυνοριακής υγείας, ε, προστασίας καταναλωτών, ποινική και αστικής δικαιοσύνης, πολιτικών δικαιωμάτων και ούτε καθεξής. και προέκυψε και η ιδέα ενός Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών, Ευρωπαϊκού Έτους Ιθαγένειας και αυτή είναι η πρώτη εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών. Αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνω σήμερα είναι μία απόπειρα να σας πω δύο λόγια για τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης η οποία έγινε για την Ιθαγένεια και όπως θα διαπιστώσετε ε, είναι πολύ ενδιαφέροντα, αποτελούν πηγή έμπνευση ε, για τις δράσεις τις οποίες ε, θέλουμε να ξεκινήσουμε ή να εφαρμόσουμε στη διάρκεια του ερχομένου έτους και νομίζω ότι το πρώτο στοιχείο το οποίο αναφέρεται από τους πολίτες όταν ρωτούνται τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μας, είναι η εμπειρία που έχουν από τη γραφειοκρατία ε, παραδείγματο χάρη όταν χρησιμοποιούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορία. Και ε, τι συμβαίνει όταν ε, ε, μεταφέρονται σε μια άλλη χώρα της Ένωσης, αναφέρονται στη γραφειοκρατία, δεν είναι σαφείς οι διαδικασίες, είναι μακρές οι διοικητικές διαδικασίες και μας λένε ε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε προς αυτό το σκοπό. Οτιδήποτε θα μπορούσαμε να κάνουμε κατά την άποψή τους σίγουρα θα αποτελέσει κάτι θετικό. Θέλουν να μειωθεί η γραφειοκρατία, για ε, ταυτότητες, ε, για άδεια παραμονής ή έγγραφα ε, ποινικού μητρώου. Αυτό λοιπόν είναι το σαφές μήνυμα το οποίο μας ε, δίνουν. Επίσης ε, λάβαμε απαντήσεις από πολίτες με αναπηρία και νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο οι πολίτες με αναπηρία να απολαμβάνουν στα άλλα κρατημέλη όλα τα ωφέλη τα οποία απολαμβάνουν ε, οι πολίτες με αναπηρία ε, και στην ε, χώρα τους. Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία μας ζήτησαν. Ένα άλλο σημείο το οποίο επισημαίνουν οι πολίτες είναι ε, το θέμα της απασχόλησης. Φυσικά αυτό δεν θα έπρεπε να εκπλήσει κανέναν. Ε, ε, βρισκόμαστε σε καιρό κρίσης. Έχουμε 25 εκατομμύρια ανέργους που αναζητούν μια θέση εργασίας και παρά το υψηλό ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού, υπάρχουν και νέες θέσεις εργασίας οι οποίες δεν ε, πληρούνται και φυσικά ε, κάτι θα πρέπει να γίνει γι' αυτό και νομίζω ότι ένα από τα στοιχεία στα οποία θα έπρεπε να επικεντρωθούμε ε, στην επόμενη έκθεση είναι ακριβώς να βοηθήσουμε τους πολίτες να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εξασφαλίσει ότι μπορούν, μπορεί κανείς να συνεχίζει να λαμβάνει για μια ε, τριμηνιαία περίοδο το επίδομα απασχόλησης, αν πηγαίνει σε μια άλλη χώρα, όμως ε, το να βρει κανείς ε, δουλειά μέσα σε τρεις μήνες δεν είναι εύκολο και η μέση χρονική περίοδος για την εξέβρεση εργασίας είναι 16 μήνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε δεν προτείνω να παρατείνουμε αυτό το επίδομα για 16 μήνες βεβαίως, αλλά νομίζω ότι μία περίοδος 6 μηνών για παράδειγμα θα επιτρέψει στους πολίτες να έχουν μια καλύτερη ε, πιθανότητα, με μεγαλύτερη πιθανότητα να βρουν ε, δουλειά σε κάποιο άλλο κρατος μέλος. Ένα ακόμα από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν ε, από τους πολίτες στην διαβούλευση είναι το θέμα της πληροφόρησης. Ο πρόεδρος τον έφερε προηγουμένως ότι είναι ελλειπή αυτή η πληροφόρηση, ενδεχομένως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην ε, το κάνει επαρκώς, ε, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα δικαίωμα των ε, πολιτών να γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν με τα δικαιώματα που έχουν. Αναφέρατε και κάποια άλλη παράμετρο, το είδαμε από το αποτέλεσμα του Ευρωβαρομέτρου ότι υπήρξε κάποια πρόοδος ε, ως προς αυτό, γιατί ένας από τους τρεις ε, πολίτες, ένας στους τρεις πολίτες ε, λένε σήμερα ότι είναι καλά ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους. Και αυτό είναι ένα ποσοστό 5% μεγαλύτερο από το 2007. Πρόκειται λοιπόν για μια σταθερή πρόοδο. Δεν ε, είναι κάτι το επαναστατικό, αλλά τέλος πάντων είναι μια καλή πρόοδος. Νομίζω ότι και το έτος ε, των, ε, του πολίτη επίσης βοήθησε σε όλη αυτή την ευαισθητοποίηση σε σχέση με τα δικαιώματα. Είναι καλό το να δημιουργούνται δικαιώματα για τους πολίτες, αλλά αν δεν τα γνωρίζουν δεν έχουν κανένα νόημα όταν γνωρίζει κανείς ε, τι να κάνει με τα ε, δικαιώματά του, το βλέπουμε και στο Ευρωβαρόμετρο, 25% ε, όσων απάντησαν είπαν ότι είναι καλά ενημερωμένοι σε σχέση με το τι μπορούν να κάνουν με τα δικαιώματά τους. 75% σημαίνει ότι δεν είναι και πάρα πολύ βέβαιοι. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να ε, δουλέψουμε περισσότερο. Δεν πρέπει απλώς να ενημερώνονται οι πολίτες για τα δικαιώματά τους. Πρέπει να τους εξηγούμε σαφέστερα, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, ότι υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν βάσει των δικαιωμάτων αυτών. Κάτι ακόμη το οποίο επίσης ε, φάνηκε στη διαβούλευση είναι τα πολιτικά δικαιώματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πλαίσιο ε, εκλογών και όσοι απάντησαν στην ε, διαβούλευση αυτή ρωτήθηκαν θεωρείτε ότι είναι φυσιολογικό να χάνετε στη χώρα σας το πολιτικό σας δικαίωμα, το δικαίωμα ψήφου σας όταν πηγαίνετε σε μια άλλη χώρα και φυσικά πάνω από δύο τρίτα απάντησαν ότι δεν θεωρούν ότι αυτό είναι σωστό. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι ε, το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει, πρέπει να ε, το δούμε πιο προσεκτικά. Το να πάει κανείς σε μια άλλη χώρα δεν σημαίνει ότι χάνει τους δεσμούς που έχει με την ε, πατρίδα του, με τη χώρα προέλευσής του. Όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, αυτό θα είναι ένα σημαντικό θέμα, είναι ευαίσθητο θέμα και θα πρέπει να το επεξεργαστούμε. Εν ολίγης, αυτά είναι κάποια από τα αποτελέσματα της ε, δημόσιας διαβούλευσης που ε, δρομολογήσαμε. Σημερινή ακρόαση είναι πολύ σημαντική για μας, γιατί είναι σημαντικό να ακούσουμε τις ιδέες σας και να τις ε, εντάξουμε στην ε, έκθεση που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9 Μαΐου. Σας εύχομαι λοιπόν μια πολύ καλή συζήτηση και ε, αναμένουμε εναγωνίως τις ε, προτάσεις που θα προκύψουν από αυτήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Λεβάιλ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, γιατί συμμετέχετε κι εσείς σε, αυτό το πάρα σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική συνάντηση για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Τις ίδιες αρχές έχουμε. Πρέπει να προσεγγίσουμε τον κόσμο να γνωρίζει ότι θα παραμείνει η Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων γιατί θεσπίζει δικαιώματα για τα 500 εκατομμύρια ε, Ευρωπαίων πολιτών, ε, ότι πρόκειται για τους πολίτες αυτούς, αυτή είναι η ε, ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετουσιώνεται σε πράξη. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις ότι όλοι οι καλεσμένοι μας εδώ στο κτίριο μπορούν να κρατήσουν την καρτούλα τα ε, ταυτοποίησης που τους δώσανε, το badge τους, και θα πρέπει να την κρατήσουν μπαίνοντα και βγαίνοντα από το κτίριο, διαφορετικά θα πρέπει να ξαναδηλωθούν και να πάρουν καινούργια καρτούλα. Στις μία η ώρα έχουμε ένα ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα, ακριβώς εδώ δίπλα, στην αίθουσα, και ε, πιστεύω ότι η συζήτησή μας θα είναι πάρα πολύ καρποφόρα και θα αρχίσουμε με το πρώτο πάνελ μας το, του οποίου συντονιστής είναι ο κ. Φιλίπ Μπουλόν, Ευρωβουλευτής και θα παρουσιάσει τους συναδέλφους μας την κυρία Κοράτσα Μπίλτ, η οποία είναι και αυτή ευρωβουλευτής, τον Μάικλ Κάσμαν, ο οποίος είναι και αυτός ευρωβουλευτής, και καλό τους συμμετέχοντες σε αυτό το πρώτο πάνελ να ανεβούν στο βήμα μαζί με τον κύριο Καμαλ Μπάρατ, συντάκτης αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Πολ Νίμιτς, ο οποίος είναι διευθυντής σε μελιό δικαιώματα και σαγένεια Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη στην Κομισιόν, και την κυρία Αντίνα Ιωάννα Βαλεάν, η οποία είναι συγγήτρια και αυτή η Ευρωβουλευτής για την έκθεση Πυρθαγιάννης Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2010 και την κυρία Άλισον Μακδόνελ από το Euro, Europa Institute Πανεπιστήμιο του Λέιντεν. Αυτή λοιπόν είναι η συμμετέχοντα στο πρώτο μας πάνελ για την επόμενη ώρα. Και το θέμα είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Και εν συνεχεία θα έχουμε την, ε, το χρόνο να ακούσουμε ερωτήσεις και απαντήσεις.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 Καλημέρα σα. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τον κύριο Λόπε Αργιλάρα, την κυρία Ρέγκμινερ και την ε, κυρία Λεμπάγια για τα εισαγωγικά του σχόλια. Σε αυτό το πάνελ θα ακούσουμε του ε, ευρωβουλευτέ, θα ακούσουμε εμπειρογνώμενε, θα ακούσουμε έναν ε, ε αναφέροντα και έναν ειδικό για τα θέματα τη Ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Θα αναφερθούμε στι δυσκολίε που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτε όταν θέλουν να ασκήσουν τα εκ των συνθήκων δικαιώματά τους ε, και θα προτείνουμε λύσεις για να μπορέσουμε να υπερβούμε τα εμπόδια αυτά. Λόγω του ότι δεν έχουμε αρκετό χώρο εδώ ε, στο Προεδρείο, κάποιοι από τους ομιλητές ε, έχουν καθίσει απέναντί μου και θα ε, λάβουν τη θέση τους εδώ στη συνέχεια. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, η Ιθαγένεια είναι μία έννοια την οποία όρισε η συνθήκη του Μάστριχτ σε υπηκόους εθνικών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ξέρω εάν πρέπει συνεχώς πώς να αντιπαραβάλουμε την εθνικότητα, ε, την υπηκότητα, συγγνώμη, με την ε, ε, ηθαγένεια διότι αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ συνδεδεμένα, γιατί η υπηκότητα βέβαια είναι κάτι το πολύ διαφορετικό από κράτος μέλος σε, κάθε, σε κράτος μέλος. η ελευθερία της κυκλοφορίας των ανθρώπων, των υπηρεσιών, των αγαθών επισυμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, μεταξύ των αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπουμε συνεχώς καταγγελίες, αναφορές, οι οποίες έχουν να κάνουν ε, με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στην άσκηση αυτής της ελευθερίας ε, μετακίνησής τους. Και έχουμε για αυτό το λόγο πάρα πολλές καταγγελίες σε σχέση με την αναγνεώρηση των επαγγελματικών προσόντων, σε σχέση με, τις, με τη διαφορετική φορολογία ή πολλές φορές πολλαπλή φορολογία, οικογενειακά οικογενειακά προβλήματα, ε, διαζύγια, συντάξεις, ε, συνταξιοδότηση, όλα αυτά έχουν, αφορούν τους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι μεταβαίνουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο για να ασκήσουν το επαγγελματικό τους, ε, την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή να ζήσουν με την οικογένειά τους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επικράτειας τα εμπόδια ε, υπάρχουν για να τα υπερβαίνουμε. Ο τρόπος για να το πετύχουμε αυτό και αυτό που μπορούμε να προτείνουμε στον ε, Ευρωπαϊκό στον Ευρωπαίο πολίτη είναι διαφόρων ειδών. Υπάρχουν οι αναφορές βεβαίως, ε, υπάρχει το δικαστήριο, ε, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει η πρωτοβουλία των ε, πολιτών από το Μάιο του 2012 που είναι ένα επιπλέον εργαλείο πλέον στη διάθεση των Ευρωπαίων πολιτών και είναι βέβαια και οι ευρωβουλευτές οι οποίοι τους εκπροσωπούν και οι οποίοι εκλέγονται από τους πολίτες. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί τρόποι έκφρασης για τους Ευρωπαίους πολίτε ε, για να μπορέσουν δηλαδή να γνωστοποιούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή του ζωή κατά την άσκηση ε, της, ε, των δικαιωμάτων τους και κατά τη διάρκεια του βίου τους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διάφοροι ομιλητές θα προσπαθήσουν να αναφερθούν στις διάφορες αυτές πτυχές ευρωπαϊκής ηθαγένειας και των προβλημάτων που προκύπτουν και μετά το πέρας των διαφόρων παρεμβάσεων θα γίνει συζήτηση στην αίθουσα ε, αυτή μέχρι ε, την ώρα ε, του γεύματος κατά τη μία η ώρα. Να μην μακρηγορήσω άλλο. Να καλωσορίσω την συνάδελφο Αντίνα Ιωάννα Βαλεάν, η συγγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκθεση περί Θαγένες Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2010 και συντονίστρια φιλελευθέρων στην Επιτροπή Αναφορών. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Θα αρχίσω λέγοντας ότι με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ να μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια που είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα από τότε που έγινα Ευρωβουλευτής το 2007. Αφορά το καθένα από εμά και όλες μας τις κοινότητες. Εγώ προέρχομαι από ένα από τα πιο καινούρια ε, κράτη-μέλη, από τη Ρουμανία και ε, έχω την εμπειρία από πρώτο χέρι πώς ε, το ευρωπαϊκό όραμα έχει βελτιώσει την κατάσταση στη χώρα μου, έχει προσφέρει νέες ευκαιρίες αλλά έχει δημιουργήσει και νέες ευθύνες. Δεν θα μιλήσω για όλα τα πλεονεκτήματα της ένταξης και της ευρωπαϊκής ιδιότητας, της ευρωπαϊκής ηθαγένειας, αλλά θα μιλήσω για πράγματα τα οποία ακόμα δυσκολεύουν τη ζωή μας. Είμαι εισηγήτρια για την έκθεση περί ηθαγένειας το 2010 και ε, παλιότερα είχα, και εισηγήτρια για την ελεύθερη κίνηση, διακίνηση πολι... συγγνώμη, ελεύθερη κίνηση πολιτών Καταρχάς λοιπόν για την ελεύθερη κυκλοφορία, ελεύθερη κυκλοφορία η οποία είναι το υπαρσμόν ε, ένα θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδρεώθηκε με την θέση ενισχύ της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία. Τα περισσότερα παράπονα ε, αφορούν το δικαίωμα εισόδου, το δικαίωμα διαμονής για πάνω από τρεις μήνες το δικαίωμα απόκτησης ε, πιστοποιητικού ε, ελεύθερης παραμονής και το δικαίωμα ε, διαβίωσης μαζί με τις οικογένειες και εισόδου μελών οικογένειας στο κράτος διαμονής. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε και έχω κουραστεί να το λέω συνέχεια να φροντίσουμε να υπερνικήσουμε και να καναργήσουμε και τα τελευταία εμπόδια από όλου ε, ε, τα τελευταία εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Και γι' αυτό χαιρετίζω με μεγάλη ικανοποίηση το έτος 2013 και την απόφαση της Κομισιόν να το ονομάσει έτος της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Εκτός λοιπόν από αυτά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ευρωπαίων πολιτών υπάρχουν και άλλα ε, εμπόδια και άλλα πολύ αρνητικά και γεγονότα τα οποία σοκάρουν. Εάν θυμόσαστε το σκάνδαλο της αποπομπής, της απέλασης ε, μελών της ε, Ρωμά, ε, της κοινότητας των Ρωμά από τη Γαλλία. Μία πράξη η οποία ήταν ντρόπια σε ολόκληρη τη χώρα και η οποία παραβιάζει κάθε διάταξη της, του δικαιώματος διαμονής και του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας. Δεν μπο, μπορούν τα επιχειρήματα ε, ε, ε, ότι κινδυνεύει η δημόσια ασφάλεια και η ένωμη τάξη να εφαρμοστούν συλλογικά πάνω σε μια συγκεκριμένη κοινότητα. Αυτά είναι θέματα τα οποία αφορούν ατομικά δικαιώματα και προσωπικές περιπτώσεις εναντίον των οποίων μπορεί να προσφύγει το κράτος. Αλλά δεν είναι δυνατον να επαναληφθεί μια τέτοια απαράδεκτη κατάσταση ξανά. Θα ε, θέλαμε λοιπόν να να σας ε, τονίσουμε ότι ορισμένες, ε, ορισμένοι, ορισμένες διατάξεις δεν εφαρμόζονται καθ' στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα παραδείγματος χάρη διατάξεις που αφορούν την συμβίωση ε, ή το, το γάμο. Ορισμένα κράτη δεν αναγνωρίζουν τη μακροχρόνια συμβίωση ω ισότιμη με το γάμο και επίσης δεν αναγνωρίζουν συμβίωση ή γάμου ομόφυλων, ε, δεν αναγνωρίζουν τα ίσα δικαιώματα με τους ετερόφιλους παρόμοιες λυπηρές διακρίσεις υπάρχουν και στην αγορά εργασίας, ε, οι τα οποία έχουν, τύχει, έχουν βγει στη δημοσιότητα. Υπάρχουν ε, ε, τόσο αρνητικά σχόλια εναντίον ε, της Βουλγαρίας και της Ρωμανίας επειδή από το 1η του 2014 θα μπορούν επιτέλους να να χαίρουν του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν, έχουν αναφερθεί στον τύπο εκατοντάδε αρνητικά σχόλια ότι θα σημειωθεί ένα κύμα μετανάστευση από τι χώρε αυτέ προ τι προς τις ε, ε, προ τι άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία είναι, είναι απαράδεκτα. Απλώ θα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τη, την ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Μάικολ Κάσμαν τώρα, μέλος της Επιτροπής Αναφερών και ε, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Είναι επίσης πρόεδρος ε, της ε, ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των λεσβιών, ομοφιλοφίλων, διεμφυλικών ατόμων. Κύριε Κάσμαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητέ Φιλίπ, ευχαριστώ σε όλους. Θα μιλήσω ελπίζω μέσα στα χρονικά μόρια, αλλά θα ήθελα να σταθώ στην ελευθερία κυκλοφορίας, στην ελευθερία διαμονής και τι γίνεται με τους θανόντες. Ένας πολύ ενδιαφέρον συνδυασμός. Θα ήθελα καταρχάς να σταθώ στο θέμα της ε, δυνατότητας πρωτοβουλίας ε, των πολιτών και το ρόλο τους στην Επιτροπή μας. Και νομίζω ότι από εκεί έχει προκύψει ακριβώς αυτό. Όταν οι πολίτες ε, συζητούν με τους ευρωβουλευτές, ασχολούμαστε με την πραγματικότητα της κατάστασής τους και ελπίζουμε ότι οι αποφασίες τις οποίες θα καταλήξουμε είναι πιο ενημερωμένες και βασίζονται περισσότερο σε λύσεις. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία χάρη χάραξης της πολιτικής και για να γνωρίζουν τι ακριβώς κάνουμε θα έχουν, πρέπει να έχουν πρόσβαση στα όλα τα έγγραφα τα οποία ε, κρατά, ε, ετοιμάζει ε, οποιοδήποτε από τα τρία θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σας μιλώ ως εισηγητής ε, του κανονισμού που κάλυπτε τα θέματα αυτά και τη αναθεώρησης και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Καπιτάνη, ο οποίος είναι εδώ σήμερα που και είναι ο πατέρας της πρόσβασης στα έγγραφα και στο ε, δικαίωμα στην ενημέρωση. Αν δεν είχε ξεκινήσει αυτός, δεν θα είχαμε αυτά τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουμε σήμερα. Για μένα η κυρία Βάλεν στάθηκε ε, και γι' αυτό και καλωσορίζω την παρέμβασή της στο θέμα της παρά... απαγόρευσης της ελευθερής κυκλοφορίας ε, οικογενειών ομοφύλων ατόμων υπάρχουν ε, κάποιοι μύθοι που κυκλοφορούν ότι επιβάλλεται ο γάμος των ομοφύλων. Ε, αυτό δεν είναι αλήθεια, δεν επιβάλλεται τίποτα στο γαμικό δίκαιο των κρατών μελών. Είναι απλώς ελευθερία κυκλοφορίας που είναι μια βασική ευρωπαϊκή αρμοδιότητα και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ε, σύμφωνα συμβίωσης και γάμοι σε άλλες χώρες θα πρέπει να καταγράφονται σε άλλες ε, χώρες όταν υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία και θα πρέπει να χαίρουν των ίδιων δικαιωμάτων που είχαν και στην ε, χώρα διαμονής τους στην προηγούμενη χώρα. Πρόκειται λοιπόν για το δικαίωμα ε, διαμονής ελευθερίας κυκλοφορίας. Αυτή τη στιγμή 8 χώρες συμπεριλαμβανομένης ε, ελπίζουμε και της Γαλλίας και του Ηνωμένου ε, Βασιλείου ε, επιτρέπουν γάμους μεταξύ ομοφύλων και επιπλέον χώρες, άλλες πέντε, επιτρέπουν και σύμφωνο συμβίωσης. Σε αυτές τις χώρες στις οποίες που υπάρχει δικαίωμα γάμου και δικαίωμα συμβίωσης, το να τους παραβιάζονται αυτά τα δικαιώματα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαράδεκτο. Να περάσω τώρα στο άλλο θέμα που θα σταθώ στην παρέμβασή μου, είναι το θέμα της, ε, του δικαιώματος ιδιοκτησίας ε, στην Ισπανία. Έχουν γίνει αναφορές ε, για το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και στο δικαίωμα της προσφυγής. Εδώ και 10 χρόνια στην Επιτροπή Αναφορών. Ε, χιλιάδες άνθρωποι έχουν πιέσει θύματα σε απάτες κτηρίων, δεν μπορούσαν να λάβουν κατάλληλη τεκμηρίωση για τα κτίρια τα οποία είχαν στην ιδιοκτησία τους, χωρίς να μπορούν να έχουν έτσι κατάλληλη ηλεκτροδότηση και ίδρυυση και έχαναν στο τέλο την κατοικία του και όλη του την αποταμίευση. Και ορισμένε φορέ ε, γινόταν κατάσχεση των οικειών του, απλώ και μόνο για λόγου αστική ανάπτυξη. Ξεκινούσε η ανάπτυξη αλλά δεν υπήρχε κανένα κέρδο για όλου αυτού του ανθρώπου. Μόνο έχαναν τα κέρδη του και είδαμε να εκδιώκονται άνθρωποι από κατοικίε τι οποίε είχαν αγοράσει νομίμω ε, να τους γίνεται έξωση χωρίς καμία αποζημίωση και ε, το πρόσχημα ήταν ε, ο Ιγιαλός. Ε, το θέμα είναι ότι αυτό το εξετάζει τώρα η Ισπανική κυβέρνηση, αλλά και εμείς ως Επιτροπή Αναφορών θέλουμε να υπάρχει δικαιοσύνη για όλους στο θέμα αυτό. Αγαπητέ Φιλίπ, ε, αν με επιτρέπει, θα ήθελα να τελειώσω σε κάτι το οποίο ίσω θα σα κάνει να μην διάσετε, αλλά είναι πολύ σοβαρό. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν ο συντονιστή μου στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ε, του έθιξε το θέμα του επαναπατρισμού των ε, θανόντων, ανθρώπων που είχαν πεθάνει σε μια ξένη χώρα και τι γίνεται με τη σωρό τους, μου είπε «Μάικολ Κάσμαν, μόνο εσύ θα μπορούσες να ξεκινήσεις να κάνεις δουλειά για πολίτες που δεν μπορούν πλέον να σε ψηφίσουν». Παρ' αυτά, το θέμα είναι θεμελιώδες. Ε, σαφώς αυτή τη στιγμή μας φορά ιδιαίτερα και θα είμαι πάρα πολύ λακωνικός. Εάν κάποιος πεθάνει αυτή τη στιγμή σε άλλη χώρα μέλος που δεν είναι η χώρα του, ε, τα εμπόδια, η γραφειοκρατία, ο πόνος ε, που θα πρέπει να υπομείνουν τα μέλη της οικογένειας σου για να μπορέσει να επανέλθει η σωρό σου στη χώρα σου, είναι δυστυχώς κάτι το οποίο πλήττει τις ζωές πάρα πολλών ανθρώπων. Ε, υπήρξα μάρτυρας ε, ενός ζευγαριού ε, που έχασαν το γιο τους ε, στις πρώτες διακοπές που έκαναν στην Ισπανία. Προσπάθησαν να μεταφέρουν τη σωρό τους, έφεραν το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους κόστισε τεράστιο ποσό χρημάτων να μπορέσουν να μεταφέρουν τη σωρό τους σε ένα μικρό φέρετρο. Το κόστος και η γραφειοκρατία ήταν τεράστια και φυσικά το άγχος και ο πόνος δεν αξίζει σε κανέναν. Δυστυχώς ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει φαίνεται ότι δεν υπάρχει, ε, υπάρχει μεν ελευθερία κυκλοφορίας μέχρι να πεθάνουμε. Και νομίζω ότι η ελευθερία κυκλοφορίας θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να μπορέσουμε να είμαστε εν τόπο χλωερό κοντά στις οικογένειές μας. Και αυτά είναι τρία σημαντικά ζητήματα τα οποία σας έθιξα σήμερα, τα οποία όπως σας είπα προηγουμένως αφορούν τους πολίτες και ξεκίνησαν από τους πολίτες. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα και όχι λιγότερα για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας που πέρασε ε, στην άλλη διάσταση κιόλα. Ε, θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο σε μία άλλη συναδελφό μας, ε, την Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ, εκ μέρους των, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Είναι επίσης εισηγήτρια για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών για τα επόμενα στάδια. Έχει το λόγο για πέντε λεπτά μετά Σήμερα το πρωί όταν ήρθα, ε, χάρηκα όλος ιδιαίτερος ε, που άρχισα την ημέρα μου στο Κοινοβούλιο συναντώντας εσάς, γιατί ο, το μεγαλύτερό μας καθήκον και η μεγαλύτερη πρόκληση είναι πώς μπορούμε να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε καθημερινά τη ζωή ε, των ε, πολιτών και να το κάνουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ είμαι μια πραγματική Ευρωπαία πολίτης. Γιατί τα λέω γαλλικά, αναρωτιέμαι, λέει η ομιλήτρια. Ε, για σένα Φιλίπ τα έλεγα στα γαλλικά τέλο πάντων. Ε, θα τα πω τώρα στα αγγλικά. Εγώ είμαι Ιταλική, Ιταλίδα, έχω Βρετανικό διαβατήριο, ζω στη Σουηδία, ε, πήρα το γαλλικό μπακαλωρέα, έχω δύο εταιρείε, είχα δύο εταιρείε πριν να εκλεγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ιταλία. εκλέγω απευθεία από του Σουηδού και έχω περάσει 30 χρόνια ζώντα σε διαφορετικά κράτη-μέλη τη Ευρωπα... της Οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ να λύσω αυτά τα προβλήματα που εκατομμύρια πολίτες ε, αντιμετωπίζουν καθημερινά, όπως και εγώ ε, προσπαθώ να ταξινομήσω ένα αυτοκίνητο ε, σε μία άλλη χώρα και να αναγνωρίσω και το, δικαίωμα, το δίπλωμα οδήγηση από άλλη χώρα που έχω. Τέλος πάντων, ε, υπάρχει έλλειψη ευαισθητοποίηση σε σχέση και με τα δικαιώματα των πολιτών αλλά και των τοπικών, ε, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάναμε πολλά πράγματα εδώ στο Κοινοβούλιο ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε στην εναρμόνιση, την καταπολέμηση της, ε, του κατακαιρματισμού, την οποία εντόπισε η πολύ καλή έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουν περισσότερα ως κοινού κανόνες, μεγαλύτερη εναρμόνιση, απλούστευση, αλλά κατά τη διάρκεια της κρίσης οι, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να υπάρχει μεγαλύτερος προστατευτισμός, μεγαλύτερη επικουρικότητα, ε, περισσότερο εθνικό πλαίσιο, το οποίο βέβαια δημιουργεί πρόβλημα σε αυτό το αίσθημα του να ανήκει κανείς σε μια κοινή ευρωπαϊκή οικογένεια. Όμω πρέπει να συνεργαστούμε γιατί η λύση της κρίσης δεν είναι λιγότερα, λιγότερη ελευθερία και περισσότερα σύνορα. Είναι περισσότερη ελευθερία. Μα το είπατε και εσείς αυτό στη διαβούλευση. Τουλάχιστον αυτό είναι το μήνυμα το οποίο πήραμε εμείς. Οπότε είμαι περήφανη που ε, είπαμε, ε, τα, είπαμε τα πράγματα όπως έχουν στην, στο πλαίσιο της οδηγίας για την προστασία των καταναλωτών. Θέσαμε τις 14 ε, ημέρες. δεν μπορώ να τα πω βέβαια όλα γιατί θα με διακόψετε κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε το θέμα ε, της προστασίας για τους άνδρες και τις γυναίκες ε, που είναι θύματα βίας, το δικαίωμα διερμηνίας, το δικαίωμα μετάφρασης, πραγματικά δικαιώματα και τα προξενικά δικαιώματα που είναι όλο και περισσότερο πρόβλημα για όσους θέλουν να ταξιδέψουν ε, ε, πρέπει να αναφερθώ και σε άλλες οδηγίες. Αν ας πούμε πάρει κανείς ένα πακέτο ταξιδιωτικό ε, σε μια άλλη χώρα, πληρώνει τα διπλά από τη στη δική σου χώρα. Όλα αυτά είναι ζητήματα για τα οποία πρέπει να συνεργαστούμε. Ο αγαπημένος μου φίλος, ε, ο κύριος Κάσμαν, θα αναφερθεί και πάλι στην πρόσβαση στα έγγραφα και θα το εμβαθύνει αυτό το θέμα ακόμη περισσότερο. Υπάρχει και το θέμα της εφαρμογής στα κράτη-μέλη, που είναι το πραγματικό πρόβλημα. Είναι πραγματικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο θέμα προστατευτισμού και βούληση, είναι θέμα τοπικής αυτοδιοίκηση ε, και καλής πίστης. Μην κάνετε τη διάκριση μεταξύ ενός Ρουμάνου, Βούλγαρου, ε, Ευρωπαίου πολίτη από άλλη χώρα που έχουν τα ίδια δικαιώματα με ε, τους ε, ε, ημεδαπούς ε, προσπαθήσαμε τόσο πολύ να σας βάλουμε ε, στη Σέγγεν και να έχετε τα δικαιώματα όλων των υπολείπων Ευρωπαίων πολιτών. Εγώ πραγματικά έχω βαρεθεί όταν μας λένε φταίνει Βρυξέλλες, όλη την ώρα Βρυξέλλες είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος. τη στην τελευταία ολομέλεια εγκρίναμε ε, νομοθέτημα που αφορά βεβαίως τους καταναλωτές. Ε, θελήσαμε όμω να δουλέψουμε περισσότερο με τα Εθνικά Κοινοβούλια και την τοπική αυτοδιοίκηση γιατί εάν η εφαρμογή ε, της νομοθεσίας δεν γίνει σωστά, μπορούμε να έχουμε την καλύτερη νομοθεσία, αλλά δεν θα δουλέψει στην πράξη. Και Φίλιπ, θα ήθελα να, τε, να ολοκληρώσω λέγοντας το εξή. Επειδή έχω ζήσει στις δύο άκρες Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ζωή μου, υπάρχει μια πραγματική πρόκληση, υπάρχει μια... Ε, κάποιο είδου δυσπιστία σε σχέση με το τι γίνεται σε μια άλλη χώρα, ότι ε, μια άλλη χώρα δεν θα μου δώσει αυτά που μου δίνει η δική μου χώρα. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε ακόμη να κάνουμε για να σπάσουμε αυτό το ταμπού, που είναι ένα πολιτιστικό ταμπού, ε, ότι η ελευθερία της ε, μετακίνησης είναι πραγματικά ένα όφελος και ότι ακόμη και ένας ασθενής, νομίζω ότι η οδηγία της ελευθερίας της μετακίνησης των ασθενών ήταν ένα τεράστιο τεράστιο επίτευγμα γιατί είναι, υπήρχαν ψυχολογικά και πολιτιστικά εμπόδια για να λειτουργήσει, να μπορεί δηλαδή ένας πολίτης να δει το όφελος αυτού του πράγματος και τώρα κάνουμε το ίδιο με τα φάρμακα γιατί δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε σε άλλη χώρα γιατί είναι διαφορετικά τα συστατικά και διαφορετικά τα ονόματα. Αν δεν τα καταφέρουμε, αν δεν κυκλοφορεί δηλαδή κανείς ε, με τα φάρμακά του στην Ευρώπη, έχει πρόβλημα να τα αγοράσει κάπου αλλού εγώ έχω ζήσει και στην Ιταλία και στη Σουηδία και θα ήθελα να σας καλέσω, έχω ψηφίσει και στις δύο χώρες και είμαι περήφανη γι' αυτό, θα ήθελα να σας καλέσω να ψηφίσετε σε ευρωεκλογέ. είμαστε συνομοθέτες, έχετε το δικαίωμα να μας ε, ε, ψηφίσετε και να μας υποχρεώσετε να κάνουμε το καθήκον μας μέσω της ψήφου σας. Ε, το... Εγώ διαφωνώ με, τις, ε, με την απόρριτη ψήφο. Κάποιος το είπε, έχετε δικαίωμα να ξέρουμε τι ψηφίζουμε, να ξέρετε τι ψηφίζουμε, για ποιο λόγο το ψηφίζουμε. Και επίσης τα κοινωνικά μίντια. Νομίζω ότι είναι ένα ε, μέρος στο οποίο συναντιόμαστε. Παρακαλούμε να μας πείτε τη γνώμη σας πάντοτε και μέσω των κοινωνικών μίντια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λίγο ξεπέρασε το χρόνο, αλλά το θέμα της επικουρικότητας το έθεσε και είναι σημαντικό αυτό, γιατί πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Οπότε, να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Καμαγίτ Μπαράτ, Βρετανό πολίτη, ο οποίος υπέβαλε ε, αναφορά σε σχέση με την οδηγία για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και των ε, οικογενειών τους για την ελεύθερη κυκλοφορία τους ε, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια σε σχέση με ανεπάρκεια προξενικών υπηρεσιών ήταν η αναφορά του. Έχετε το λόγο, κύριε Μπαράτ, για 10 λεπτά. Καταρχάς ευχαριστώ τους ε, οργανωτές ε, σήμερα για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης. Θέλω να τονίσω τρία σημεία τα οποία συνδέονται με την επαγγελματική και προσωπική μου ζωή. Όταν αναγκάστηκα να υποβάλω αίτηση για βίζα Schengen. Θα αναφερθώ λοιπόν καταρχάς στα προβλήματα που είχα όταν ζήτησα τη μία θεώρηση, μία βίζα για τη γυναίκα μου η οποία ήταν Ινδύ υπήκος. Δεύτερο, τα προσκόμματα που είχα ως φοιτητή και τρίτον, ε, για το ρόλο της τοπικής αυτοδείξης. γιατί εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλο και δουλεύω <clears throat> για την τοπική αυτοδείξη στην περιφέρεια μου. Πιο κοντά στο μικρόφωνο παρακαλώ. Λοιπόν, ε, ως σαν οικογένεια αποφασίσαμε να κάνουμε τις διακοπές μας, να εκμεταλλευτούμε ε, μια προσφορά διακοπών και η γυναίκα μου είχε ειδικό διαβατήριο και χρειαζόταν να πάρει μία θεώρηση, μία βίζα. Και κάναμε λοιπόν μία έρευνα, αν θέλετε, για να δούμε τι χρειάζεται να υποβάλουμε για τις διάφορες θεωρήσεις στα διάφορα μέρη του κόσμου. Από τις προφορίες που σύλλεξαμε το πράγμα φαινόταν απλό. Όμως η θεωρία δεν, ήταν, ε, η θεωρία δεν μεταφραζόταν στην πρακτική καθόλου. οι περισσότερες χώρες σε παραπέμπουν σε, μια άλλη, σε έναν άλλο πράκτορα που ασχολείται με τις ε, βίζες και πραγματικά ε, έχουν αναθέσει λοιπόν σε εξωτερικές υπηρεσίες και πρακτορία ε, τα δικαιολογητικά και την όλη διαδικασία των θεωρήσεων, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά απογοητευτικό. Χρειάζεται παραδείγματο χάρη να αποδείξεις τι ε, τραπεζικούς λογαριασμούς έχεις. Χρειαζόταν η άδεια οδήγησης και αυτό το οποίο ε, με υποχρέωσε και το βρίσκω παράδεικτο είναι ότι χρειάζεται να πληρώσω χαράτσι επιπλέον και επίσης ε, μπορούν να χειριστούν μόνο 60 ε, άτομα, 60 αιτήσει ε, θεωρήσεων την ημέρα. Άρα λοιπόν, για να προχωρήσεις σε αυτή την αίτηση πρέπει να σηκωθεί μέσα στην άγρια νύχτα, να πας να στηθείς στην ουρά τα χαράματα στο προξενείο για να μπορέσεις να πάρεις τα δικαιολογητικά και εν συνεχεία να πας στο πρακτορείο κλπ. κλπ. Και τελικά ε, σκέφτεσαι θα με πάρουν σήμερα, είμαι μέσα στους 60 των οποίων την αίτηση θα εξετάσουν ή είμαι ο 61ος και θα με διώξουν για να ξανάρθω αύριο. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μετρούσαν πόσοι ήταν στην ουρά. Προσπάθησα να εξηγήσω ότι κάνω την αίτηση θεώρησης κάτω υπό τη διαδικασία της ελεύθερης κυκλοφορίας και παρόλα αυτά αναγκάστηκα να υποβάλω γράμματα από τον εργοδότη της, ε, τα τραπεζικά έγγραφα, το δίπλωμα οδήγησης, ε, το, την άδεια κυκλοφορία του αυτοκινήτου που δεν καταλαβαίνω καθόλου τι σχέση είχε. Δεν είχα δηλαδή καμία επιλογή παρά να υποβάλω όλα αυτά τα δικαιολογητικά. Αναγκάστηκα να πάρω μία ημέρα άδεια από τη δουλειά μου για να τα κάνω όλα αυτά. Μάζεψα λοιπόν ένα μάτσο χαρτιά και τους τα έδωσα. Λέω πάρτε τα και κάντε καλά. Γυρνώντας λοιπόν πίσω στο σπίτι μου με το τρένο σκεφτόμουν τι γίνεται εδώ και έστειλα ένα email, ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στον Ευρωβουλευτή της Περιφέρειας μου. Περίμενα δύο εβδομάδες, χαίρομαι που δεν ήταν κανένας από εσά και εσείς κύριε Κάσμαν. Δύο εβδομάδες δεν είχα καμία απάντηση και είπα ότι ε, κάτι επιτέλους πρέπει να κάνω. Μπήκα πάλι στο διαδίκτυο, κοίταξα την πληροφόρηση που υπάρχει εκεί, ξαναεξέτασα όλη τη διαδικασία για τις θεωρήσεις. Συγγνώμη, ε, ε, έχω λίγο τρακ γιατί δεν είμαι συνηθισμένο να μιλάω έτσι σε ακροατήριο. Εν πάση περιπτώσει, εξέτασα όλη τη διαδικασία, όλες τις διατάξεις, επίσης τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων. και διαπίστωσα ότι ε, τα πράγματα είχαν λίγο προχωρήσει περαιτέρω, διότι υπάρχει και διαδικασία κύρωσης αν δεν τηρηθούν οι διαδικασίες. Και είδα ότι το προξενείο δέχεται τώρα αιτήσει με ραντεβού. Πρέπει να κλείσει δηλαδή ένα ραντεβού, αλλά και πάλι σε πιέζουν να πα στο πρακτορείο για να πληρώσει το χαράτσι. Δηλαδή σου λένε, ναι, μεν θα χειριστούμε εμεί την αίτησή σου, ε, η οποία θα κάνει χήμερες, αλλά αν θέλει να τελειώνει γρήγορα πήγαινε στο μπράκτορα τάδε και αυτό θα τα διευθετήσει πιο γρήγορα. Γίνεται λοιπόν αυτό το πρακτορείο δεν ε, το ενδιαφέρει καθόλου αν εσύ είσαι Ευρωπαίος πολίτης ή όχι. Σε βλέπει σαν νούμερο πελάτη και σε ε, διαχειρίζεται, σε μεταχειρίζεται σαν το πελάτη Χ ποσό τον ενδιαφέρει αν είσαι Ευρωπαίος ε, πολίτης ε, ή έχει ευρωπαϊκή εισαγένεια ή όχι. Ξανά λοιπόν πήγα στο διαδίκτυο και στην ελεύθερη κυκλοφορία και το... οι πληροφορίες για την ελεύθερη κυκλοφορία είχαν ένα τμήμα που αναφερόταν στις θεωρήσεις. Το έγγραφο αυτό όταν το πάτησα ήταν σε format PDF 47 σελίδες. 47 σελίδες. Είναι δυνατόν ένας Ευρωπαίος πολίτης να διαβάσει 47 σελίδες για να δει ποια είναι τα δικαιώματά του. Εάν έχεις πάει στη νομική σχολή και είσαι νομικός, ενδεχομένως. Αλλά αν είσαι απλός πολίτης, πώς είναι δυνατόν. Υπάρχει λοιπόν ένα, μια άλλη παραπομπή στα 47 47 αυτές σελίδες για τους Ευρωπαίους πολίτες. Πατάς λοιπόν σε, αυτή την, ε, σε αυτό το σύνδεσμο και έχει άλλο ένα σωρό εγγράφων με περίπλοκες πληροφορίες ε, και διατάξεις για το πώς θα χειριστείς αυτό το θέμα. Εν μεταξύ, ε, είχαμε στεναχωρηθεί, είχαμε συγχυστεί, τέλος πάντων αυτές οι διακοπές μας βγήκαν από τη μύτη την επόμενη χρονιά αποφασίσαμε να πάμε στο Άμστερνταμ. Πήγαμε, ε, πήγα πάλι στην ιστοσελίδα της ε, ε, πρεσβείας και πολύ γρήγορα είχαμε μία απάντηση τι χρειάζεται. Πήγα στο προξενείο στο Birmingham, στο Ολλανδικό προξενείο στο Birmingham και μέσα σε 72 ώρες είχαμε τη βίζα της γυναίκας μου, τσάκα τσάκα, όλα πήγανε πολύ ομαλά και ε, διαπίστωσα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις και για ορισμένες χώρες τα πράγματα δουλεύουν ρολό και σε ορισμένες άλλες δεν δουλεύουν καθόλου. Αυτά όσον αφορά την ταλαιπωρία μας για τις θεωρήσεις. Το δεύτερο μου σημείο αφορά Α, αφορά το γυμνάσιο, το Λύκειο της περιφέρειάς μου, όπου ήμουνα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ε, του σχολείου αυτού. Και ε, είχα μία συνάντηση με την υπεύθυνο για ε, τους μαθητές του Λυκείου, δηλαδή τους άνω των 16 ετών. Στην Αγγλία έτσι υπάρχει αυτή, αυτή ας πούμε ο διαχωρισμός και μετά τα παιδιά αυτά πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Και ήθελα να διευκρινίσω ορισμένα θέματα για σπουδές στο εξωτερικό, εκτός Ηνωμένου Βασιλείου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μην ξεχνάτε παρακαλώ ότι έχουν ανεβεί τα δίδακτρα τώρα για τα πανεπιστήμια για την τριτοβάσμια εκπαίδευση στις 9.000 λίρες κατά μέσο όρο. Οπότε ενδιαφέρονται πάρα πολλά παιδιά και γονείς εάν υπάρχουν φθηνότερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη να πάνε εκεί. Όμως κανένα παιδί, κανένας μαθητής ε, του Λυκείου δεν είχε υπόψη του ότι έχει αυτό το δικαίωμα να σπουδάσει αλλού. Κανένας δεν είχαν ε, χαμπάρι όπως λέμε. Ε, τα παιδιά αυτά δεν ξέρανε πού να ψάξουν, πώς να ψάξουν. Βεβαίως, όταν περνάνε από τάξη σε τάξη, έχουν ε, μάθημα για τα δικαιώματα του πολίτη, δεχομένως και κάποιες συμβουλές για την επαγγελματική τους καρτάστηση κλπ. Αλλά με την εχθρότητα που υπάρχει στα, στο βρετανικό τύπο κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά είναι συνήθως στο σκοτάδι για τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό πρέπει να τα πλησιάσουμε αυτά τα παιδιά, αυτούς τους σπουδαστέ και να τους πούμε «Κοιτάξτε, έχετε αυτά τα δικαιώματα και μπορείτε να πάτε ελεύθερη κυκλοφορία». Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο εμπόδιο και ο συνήθως είναι οικονομικό. Τα χρήματα τα οποία παίρνουν για τις σπουδέ τους καταβάλλονται από την κυβέρνηση μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης και δεν είναι υποτροφία, είναι δάνειο. Τα, τα χρήματα αυτά λοιπόν που παίρνουν είναι δάνεια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα οποία βεβαίως θα αποπληρώσουν συνεχεία στην κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σπουδαστές οι μαθητέ που προέρχονται από τι πιο φτωχέ περιοχέ, ούτε καν ε, δεν έχουν καμία ευκαιρία να εκμεταλλευτούν αυτέ τι δυνατότητε να σπουδάσουν στο εξωτερικό, να ζητήσουν τα χρήματα αυτά από τη Βρετανική κυβέρνηση διότι δεν έχουν αυτή η κυβέρνηση, δεν τους επιδίνει αυτή τη δυνατότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν δεν έχεις κάποια υποτροφία ή εικονιακά μέσα, δεν μπορείς να εκμεταλλευτείς αυτή τη δυνατότητα τα, εμείς θέλουμε τα παιδιά αυτά να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δάνεια, αυτά τα κονδύλια που παίρνουν ε, για να με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως νομίζουν ότι είναι καλύτερο για τις σπουδέ τους. Όμως αυτό δεν γίνεται. Υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία νε, νεότητα σε, σε κίνηση. Ε, είναι μια πρωτοβουλία μέσω της οποίας μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το 20% που μετακινείται από την νεολαία, από το νέο πληθυσμό, είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού μας. Δεν προέρχεται μόνο από μια κοινωνική τάξη, αλλά αντιπροσωπεύει όλες τις κοινωνικές τάξεις. Δεν είναι μόνο από οικογένειες που έχουν τα εισοδήματα και μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία, αλλά ότι προέρχονται και από τις πιο στερημένες, ε, στε, στε, στερημένα στρώματα του πληθυσμού στην Επιτροπή των πληροφοριών, πληροφοριών μιλάνε συνέχεια για την ενημέρωση, τη συνειδητοποίηση τι γίνεται σε τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ δουλεύω ε, για το Δήμο της περιοχής μου και όταν ένας κάτοικος της περιφέρειας μου του Warwickshire ήθελε να ξέρει ποιος, ε, ε, ποιος είναι υπεύθυνο για το φωτισμό ή για τα σκουπίδια της περιοχής μου, είχε τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε, τρία διαφορετικά, ε, σε τρεις διαφορετικές διευθύνσεις του Δήμου. Αυτό ήταν περίπλοκο διότι ο ένας τον, ε, το, του έριχνε, τον μπαλάκι στον άλλον για τις πληροφορίες. Τώρα τα ορθολογήσαμε όλες αυτές τις υπηρεσίες και έχουμε ένα κομβικό σημείο όπου ο πολίτης μπορεί να απευθυνθεί, ο δημότης δηλαδή, και να πάρει τις πληροφορίες που θέλει. Από ένα σημείο, μία διεύθυνση ένα άτομο. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να ορθολογιστούν, πρέπει να βελτιωθούν έτσι ώστε οι τοπικές κοινότητες και οι δήμοι να μπορούν να ενσωματώσουν αυτές τις προφορίες και να τις διοχετεύσουν περαιτέρω στους ενδιαφερόμενους. Είναι ο καλύτερος τρόπος να ε, διανύμουμε τις πληροφορίες και να ενημερώνουμε τους πολίτες μας μέσω του Δήμου, μέσω της τοπικής ε, αυτοδιοίκησης. Αντίθετα όμως, τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Δήμοι κατηγορούν συνέχεια και εκφράζονται εχθρικά κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα το οποίο δημιουργεί όλα αυτά τα προσκόμματα. Αυτά είχα να πω. Ε, Γενικώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαράκ, για αυτή τη μαρτυρία σας. Σας έδωσα λίγο περισσότερο χρόνο διότι δεν είστε μαθημένος όπως οι ευρωβουλευτές να μιλούν μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Υπήρχε και το συγκινησιακό κομμάτι το οποίο ε, μας παρουσιάσετε σήμερα και πραγματικά όλα όσα μας είπατε είναι... Ε, ε, εγγεγραμμένα στην καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Αναφερθήκατε στις διάφορες διατάξεις που έχει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσει την παιδεία, την ανταλλαγή, την ανώτατη εκπαίδευση από τη μία χώρα στην άλλη. Πρόκειται για διατάξεις οι οποίες ε, είναι πολύ αποτελεσματικές και λογικά θα έπρεπε να επιτρέπουν στους νέους στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια να μπορούν να αποκτήσουν αυτή την ευρωπαϊκή θα γένεια, αυτή την έννοια του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σταθήκατε και στα διοικητικά προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν στη συνέχεια στην καθημερινότητά του με τις διοικητικέ υπηρεσίες που ε, ουσιαστικά τους καθυστερούν και μόνον. Πρέπει λοιπόν να καλύψουμε όλο αυτό το φάσμα. Ε, υπάρχουν και τα θέματα των μέσων μαζική ενημέρωσης, τα οποία αναφερθήκατε δεν έχουμε μόνο τα εθνικά μέσα μαζική ενημέρωση, αλλά και τοπικά μέσα ενημέρωση, τα οποία δυσκολεύονται ορισμένε φορές να κατανοήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μεταδίδουν μέχρι τον πολίτη εκεί στον τόπο του τι ακριβώς του προσφέρει η Ευρώπη. Θα επανέλθουμε βέβαια στα όσα μας είπατε στη συνέχεια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μαρτυρία σας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Τόνι ε, Βενάμπλε, Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Δράσης των Πολιτών ε, και ασχολείται με θέματα ελεύθερης κυκλοφορίας, δικαιωμάτων των πολιτών και προστασίας των καταναλωτών στην Ευρώπη. Μετά από την παρουσίαση αυτή θα ακούσουμε τον κύριο Τόνι Μακουίν, Γενικό Διευθυντή του Ιρλανδικού Διοικητικού Συμβουλίου Πληροφοριών. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μακουίν είναι εδώ. Α, συγγνώμη, ναι. πριν ο κύριος ε, Μακουίν ήταν ε, ε, Γενικός Διευθυντής Κοινωνικών Υπηρεσιών και Πληροφοριών. Να δώσω πρώτα τον λόγο στον κύριο Βενάμπλ για ένα τέταρτο περίπου, δεν ξέρω πότε πρέπει να φύγετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε να πω κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με τα όσα μόλις ακούσαμε από τον αναφέροντα, διότι εμείς δίνουμε συμβουλές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε μια ομάδα 60 νομικών εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται πλέον με 17.000 ερωτήματα ετησίως, ε, τα οποία γίνονται όλο ένα και πιο περίπλοκα. Και από αυτά τα ερωτήματα πολλά έχουν σχέση με τα όσα ε, αναφέρουν συχνά οι πολίτες ε, και για την οδηγία 2004-38, την οδηγία για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, ένα 50% ε, είναι ιδιαίτερα προβληματικά, θα μπορούσα να πω, και μπορούν να οδηγήσουν σε διαδικασίες επί παραβάση και είναι πολύ πιο περίπλοκη και σύνθετη διαδικασία επίλυσής τους. Προσφάτως ε, συστήσαμε μία ε, κλινική ευρωπαϊκών δικαιωμάτων, η Rights Clinic, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πιο ακαθόδη ζητήματα σε συνεργασία με μη κυβερνητικέ οργανώσεις πανευρωπαϊκά, διότι βλέπουμε ότι ε, φθήνει ο σεβασμός των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων στον οποίο αναφερθήκαμε. Και πολύ εύστοχα το ανέφεραν όλοι αυτό. Αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω εγώ είναι ε, το εξής. Γιατί χάνουμε το δάσος και βλέπουμε μόνο τα δέντρα. Φέτος που έχουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών, αυτό που θα θέλαμε είναι μία χάρτα. Μία χάρτα την οποία χρειαζόμαστε για τέσσερις λόγους. Καταρχάς, διότι κανείς δεν γνωρίζει στην πραγματικότητα τι περιλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια υπάρχει μια μεγάλη αναγνώριση ως ονομασία, αλλά αν κάποιος αναζητήσει λίγο βαθύτερα και προσπαθήσει να κατανοήσει τι θεωρούν οι πολίτες ότι είναι, ακόμα και αυτό το 25% που διαβάζει παραπέρα από τις ετικέτες, οι απαντήσεις είναι μάλλον ασαφείς. Βρισκόμαστε λοιπόν ενώπιον μιας κατάστασης όπου όλοι γνωρίζουν ε, τι είναι ένα ε, προπαρασκευασμένο κατεψυγμένο γεύμα, αλλά δεν γνωρίζουμε από πού προέρχεται και τι περιλαμβάνει. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση λοιπόν που θα μπορέσει να επιλύσει το πρόβλημα αυτό από μόνο του. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε μια χάρτα είναι διότι χρειαζόμαστε περισσότερη συνέργεια σε θεσμικό επίπεδο. Έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος ε, με την ε, ενιαία θηρίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πληροφορίες και συμβουλές, αλλά το νομοθετικό πλαίσιο εξακολουθεί να εμπίπτει σε διάφορες αρμοδιότητες, διάφορες γενικές διευθύνσεις και οι διάφορες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιλαμβάνονται διαφορετικά την ευρωπαϊκή ηθαγένεια, ενώ θα πρέπει στην πραγματικότητα να υπάρχει ένα οργανωμένο πλαίσιο. Ο τρίτος λόγος που έχει σχέση και με το προηγούμενο είναι ότι λόγω του κατακαιρματισμού και εντός των θεσμικών οργάνων είναι πάρα πολύ δύσκολο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργηθεί ε, μια ε, κοινωνία των πολιτών ε, περιφερειακό επίπεδο που θα μπορέσει να αποτελέσει την όθηση. Και το ίδιο ισχύει και για το ακαδημαϊκό έργο. Πέραν των νομικών, των πολιτικών επιστημόνων, κοινωνιολόγων και φιλοσόφων που θα έπρεπε κανονικά να συνεργαστούν σε ένα ε, οργανωμένο πλαίσιο, ο καθένας εργάζεται μεμονωμένα στο ε, κλουβάκι του και Τελικώς η ευρωπαϊκή ηθαγένεια μπορεί να είναι απλώς ε, μια αφαιρημένη έννοια την, η οποία θα άγεται και φέρεται προς διαφορετικές καθεστήσεις ανάλογα με τα συμφέροντα του καθενός. Ελπίζουμε λοιπόν να υπάρξει αυτή η χάρτα σε αυτό το ευρωπαϊκό έτος. Και τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η χάρτα. Το εφαλτήριο, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να είναι το δικαίωμα στην ενημέρωση των πολιτών, να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους, τι μέσα πρόσβασης έχουν προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και πώς μπορούν να συμμετέχουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο ως ε, δραστήριοι Ευρωπαίοι πολίτες. Ετοιμάζουμε λοιπόν, καταρτίζουμε αυτή τη χάρτα ε, με βάση αυτές τις τρεις συνιστώσεις ε, ε, των δικαιωμάτων, της πρόσβασης και το δικαίωμα του ανήκειν. Θα ήθελα να πω το εξή. Ε, όταν ξεκινάει η διαδικασία, αντιλαμβάνεσαι ότι ο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι πολίτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ περιορισμένο. Ε, είναι πολύ ευρύτερο το πλαίσιο από τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Είναι το ευρύτερο πλαίσιο τη έλλειψη διακρίσεων, όχι μόνο για του πολίτε ε, που μετακινούνται και κυκλοφορούν, αλλά και για του πολίτε που διαμένουν μόνιμα κάπου. Για να μπορέσουμε λοιπόν να αντιληφθούμε ποια είναι η ευρωπαϊκή ηθαγένεια, θα πρέπει να προσθεθούν πολύ περισσότερα στοιχεία. Και θα ήθελα να ε, κάνω τρεις παρατηρήσεις για αυτές τις τρεις συνιστώσεις, πολύ σύντομα και θα πρέπει να με διακόψετε εδάλλως κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, για τα δικαιώματα. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι το κυρίω θέμα για τη χάρτα δεν είναι να επινοήσουμε νέα δικαιώματα, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα υφιστάμενα ε, έχουμε μια νέα εκδοχή μιας ε, παλαιότερης έκθεσης με τίτλο Mind the Gap για την καλύτερη εφαρμογή των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων. Δεν θεωρούμε ότι συντρέχει κάποιος λόγος, αυτή τη στιγμή που έχουμε τη χάρτα, ε, να πρέπει να έχει Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για την προστασία μιας επιχείρησης κατά του αθέμητου ανταγωνισμού ε, και όχι για την εφαρμογή των ε, ευρωπαϊκών δικαιωμάτων. Θα πρέπει λοιπόν το σκεπτικό μας να είναι να εφαρμόζεται σωστά, να εφαρμόζεται γρήγορα και να υπάρχει προληπτική δράση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εδώ θα κάνουμε προτάσεις ε, στη χάρτα. Το δεύτερο θέμα που αφορά την πρόσβαση είναι ότι ναι, συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος ε, και να υπάρχει πρόσβαση σε έγγραφα ώστε να είναι πιο αυθεντική αυτή η ελευθερία ενημέρωσης ε, και όπως και ο αναφέρον δίνουμε και εμείς μια μάχη και για μας είναι οργανωμένο το λόμπι εδώ, δεν είναι εύκολα τα πράγματα Τόσα χρόνια ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγγραφα τα οποία σχετίζονται με την δυνατότητα opt-out από τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής στάθηκε στο πλευρό μας και εξέδωσε μια πολύ επικριτική σύσταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του Ετου και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα δίνει πλήρη πρόσβαση στις ε, νομικές ε, γνωμοδοτήσεις ε, για τη δυνατότητα opt-out του Ηνωμένου Βασιλείου, της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Πολωνίας από τη Χάρτα. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια ένδειξη διαφάνειας από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι σωστό για μια κυβέρνηση να αναφέρεται στη δημοκρατία στη χώρα της και από εκεί και πέρα να αναμένει ότι όλα θα είναι απολύτως απόρριτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βέβαια αυτή η μάχη είναι πάρα πολύ μεγάλη και δυστυχώς ε, μακρηγορεί πάρα πολύ και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για νίκη. Αλλά ε, μας ενδιαφέρει ε, να υπάρχει κάθε μορφής πρόσβαση στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφοράες, ε, συστάσεις, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία κατά την άποψή μας δεν χρησιμοποιούνται επαρκείς και δεν είναι απόλυτα ασφαλείς αυτοί οι μηχανισμοί. Ε, κατόπιν θα δούμε αυτή την αίσθηση του ανήκει, του να ανήκει κάποιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με το, δυνατότητα του ενός εκατομμυρίου υπογραφών ε, της ε, πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων ε, πολιτών. αρχίζει να χρησιμοποιείται, ο κόσμος αρχίζει να επιτυγχάνει τους στόχους τους. Γιατί λοιπόν να μην μπορούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, πιο ακριβείς και σε άλλες πτυχές της συμμετοχικής δημοκρατίας βάσει του άρθρου 11 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πιο ευρωπαϊκές ευρωεκλογές ε, με υπερεθνικές λίστες για παράδειγμα. Υπάρχουν μια σειρά από αλλαγές που θα μπορούσαμε να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν καταρτίζουμε ε, αυτή την έκθεση. Θέλουμε να την ε, ε, δημοσιεύσουμε για ευρύτερη συζήτηση το συντομότερο δυνατόν και ελπίζουμε ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι απόψεις μας από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ιδίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι εκεί νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ελπίδα προόδου αυτής της ιδέας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Δεν για την πρότασή σας για τη χάρτα. Θα τη λάβουμε σοβαρά υπόψη. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μακουίν. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, είμαι πολύ ευτυχής που έχω την ευκαιρία σήμερα να μιλήσω για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Έχω μία παρουσίαση με διαφάνεια, την οποία δεν θα παρουσιάσω διότι είναι πάρα πολύ πυκνή, αλλά θα ήθελα να επικεντρώσω την προσοχή σας στη δεύτερη διαφάνεια η οποία δείχνει τις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια και το βαθμό στον οποίο οι Ευρωπαίοι πολίτες μετακινούνται μέσα στην επικράτεια. Έχουν μετακινηθεί δηλαδή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ε, Επικράτειας. Όμως στην Ιρλανδία η κατάσταση είναι διαφορετική. Έχουμε δει 4,5 εκατομμύρια είναι ο πληθυσμό στην τελευταία απογραφή της Ιρλανδίας. Τα τελευταία 20 χρόνια και ειδικότερα τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε δει μια τεράστια μετανάστευση από άλλα μέρη της Ευρώπης ε, στην Ιρλανδία και τώρα 12% του Ιρλανδικού πληθυσμού είναι μη Ιρλανδοί ε, δηλαδή 450.000 άτομα περίπου, 366.000 άτομα ε, είναι ε, Ευρωπαίοι πολίτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Πολωνία, από τη Λιθουανία, από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και αυτό βέβαια έχει πάρα πολύ ε, σημαντικό αντίκτυπο και θετικό αντίκτυπο και ειδικότερα στην κατάσταση στην Ιρλανδία. Αυτό έγινε σε μία περίοδο ανάπτυξης ε, στην Ιρλανδία από το, 2010, από το 2007. Όταν περάσαμε αυτό το σκόπελο 2007-2008 είδαμε ότι αυξήθηκε η μετανάστευση ε, ενώ η μετανάστευση από την Ιρλανδία δεν είναι μεγάλη. Είναι γύρω στα 87.000 άτομα. Πολύ περισσότεροι έρχονται όμως στην Ιρλανδία Ιρλανδία. Επομένως έχουμε μια πολύ ε, μεγάλη ε, εμπειρία σε μικρό χρονικό διάστημα από τον αντίκτυπο της μετανάστευση. Εμείς υποστηρίζουμε μη κυβερνητικέ οργανώσεις, υπηρεσίες πολιτών ε, για να βοηθήσουμε ε, τους ανθρώπους αυτούς. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη πείρα από ανθρώπους που έρχονται στην Ιρλανδία και έχουν προ, θέλουν να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματά τους, θέλουν να ενημερωθούν για τα δικαιώματα αυτά. Το 2012 για παράδειγμα είχαμε πάνω από 600.000 ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενημέρωσης των πολιτών, 10-11% από αυτούς, δηλαδή 60 με 70.000 άτομα περίπου, είναι άνθρωποι που είναι ε, Ευρωπαίοι πολίτες έχουν έρθει τις περισσότερες περιπτώσεις να δουλέψουν στην Ιρλανδία και ζητούν πληροφορίες για τα δικαιώματά τους. Ε, η ανεργία είναι περίπου 14% στην Ιρλανδία αυτή τη στιγμή. Μεταξύ των μη Ιρλανδών είναι υψηλότερη, είναι 18%. Οπότε αυτό έχει να κάνει βέβαια με αύξηση των ε, ετοιμάτων σε σχέση με τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Υπήρχαν όμως και πολλά θέματα που αφορούσαν τα δικαιώματα δικαιώματα απασχόληση από το 2008 και μετά, όμως είναι περισσότερο δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης. Ε, το, τα θέματα λοιπόν που προκύπτουν για μας είναι πρόσβαση στις υπηρεσίες, χρήση γλωσσών, ε, άνθρωποι προσπαθούν να καταλάβουν ε, τις διάφορες θεσμικές δομές που είναι διαφορετικές από αυτές που γνωρίζουν από τη χώρα τους, ε, τρόπους αντιμετώπισης των κυβερνητικών υπηρεσιών και προβλήματα βέβαια εφαρμογής. Κατά την άποψή μας η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας είναι πάρα πολύ σημαντική. Είχε πάρα πολύ θετικό αντίκτυπο στην Ιρλανδία κατά τα τελευταία 40 ε, χρόνια όσον αφορά τη μεταγραφή των δικαιωμάτων απασχόλησης που χρησιμοποιούνται σε άλλα μέρη της Ευρώπης, ε, δικαιώματα ε, ισότητας, δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης. Είχαν πάρα πολύ θετικό αντίκτυπο του τουλεχθέντος Υπάρχουν, υπάρχει είναι διαφορετική κατάσταση στην Ιρλανδία. Ε, το να μπορέσει κανείς ε, να ενσωματώσει το, ε, την ε, ιδέα της ευρωπαϊκής ηθαγένειας είναι πολύ σημαντικό. Αν μένει κανείς στο Δουβλίνο ή στη Δυτική Ιρλανδία, ε, νιώθει κανείς Ιρλανδός, αλλά δεν καταλαβαίνει πολύ καλά, δεν νιώθει, πολύ καλά, δεν νιώθει πάρα πολύ Ευρωπαίος. Αν καταλάβει όμως καλύτερα τι εκπροσωπούν οι Βρυξέλλες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αλλάξουν τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωση των ε, Πολιτών ε, προσπαθεί να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό. Και θα ήθελα να παραθέσω κάτι που νομίζω ότι έχει ε, σημασία. Ο Brian Brewer που ήταν Αυστραλός ε, είπε ότι όσον αφορά την, ε, τις καταγγελίες, τις προσφυγές είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο μέσος πολίτης συνήθως βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Οι δημόσιες υπηρεσίες έναντι των οποίων μπορεί να γίνονται καταγγελίες μπορεί να έχουν καλύτερο στάτους, καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες και καταλαβαίνουν καλύτερα τις πολιτικές και τις διαδικασίες. Επομένως, ε, ε, οι πρωτοβουλίες υπέρ των πολιτών εξισορροπούν κάπως το σύστημα και το καθιστούν δικαιότερο. Έχοντας λοιπόν αυτό υπόψη μας σε σχέση με την επικουρικότητα και σε σχέση με την κατανόηση των προβλημάτων που υπάρχουν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη πρακτική και στο πλαίσιο των Βρυξελών και στο πλαίσιο των εθνικών ε, θεσμών. Οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την νομοθεσία, για τους κανόνες ε, και που εργάζονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, πρέπει να έχουν την πείρα της πραγματικής μεταχείρισης των καταγγελιών κάθε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μαρτυρία σας, την Ιρλανδική σας μαρτυρία. Θα ήθελα τώρα να καλέσω την Άλισον Μακδόνελ ε, από το Europa Institute, Πανεπιστήμιο του Λάιδεν, συνεκδότρια της επιθεώρησης Common Market Law ε, που ενδιαφέρεται για το ευρωπαϊκό ε, δίκαιο σε γενικές γραμμές, να μας μιλήσει για κάποια σημαντικά ζητήματα, ε, την ηθαγένεια και, την, και διάφορα νομικά ζητήματα. Έχετε 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ και για μένα είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκουμε εδώ σήμερα. Εγώ θα προσδώσω μια πιο, ένα πιο ακαδημαϊκό τόνο στη συζήτηση και ελπίζω να μην έχετε την άμεση αντίδραση ότι αφού είναι ακαδημαϊκό δεν με ενδιαφέρει ή δεν με αφορά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα δεδομένου ότι ε, συνήθως εξετάζουμε περιπτώσεις που προκύπτουν και οι οποίες περιπτώσεις απαιτούν μία εξέβρεση λύσεως. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν ε, στην τεκμηρίωση του τομέα μου Έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις και αναλύσεις περιπτώσεων. Οι περισσότερες αφορούν ονόματα. Ονόματα. Πώς δημιουργούνται και πώς γράφονται. Πολλά χρόνια υπήρχε αυτό το ζήτημα πριν από τις καινούργιες εξελίξεις που αφορούν την Ιθαγένεια και την κυκλοφορία. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό νομίζω γενικά για την ομολογία που έχει σχέση με τα ονόματα είναι ο τρόπος με τον οποίο διαφαίνεται η ανάγκη εξέβρισης μιας ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων μεμονωμένων πολιτών να διαλέξουν πώς, πώς θέλουν να εκφράσουν και να γράψουν το όνομά τους ιδίως ε, διασυνοριακά, Παραδείγματο χάρη όταν γεννιέται το παιδί του, ή όταν παντρεύονται. Ε, προκύπτουν μεγάλα ε, γραφειοκρατικά προβλήματα όταν χώρες έχουν με διαφορετικές διαδικασίες και διαφορετική κουλτούρα και απαιτεί διατάξεις. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ όλων αυτών των διαδικασιών, δεδομένου ότι μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει να διαφυλαχθεί και η εθνική ιδιότητα και η πολιτισμική διά, ε, διάσταση των πολιτών. Δηλαδή, ε, έχει άμεση σχέση η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη και με τον καταστατικό χάρτη, τον, τους εθνικούς καταστατικούς χάρτες, αλλά και με την ομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο επέτρεψε ε, στο Αυστριακό κράτος να επιβάλλει τις ε, διατάξεις του όσον αφορά τις, ε, τους κανόνες γραφής και ιδιότητος ενός ονόματος. Ο δεύτερος τομέας, ε, ο οποίος ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, είναι η εναρμόνιση του ιδιωτικού δικαίου. Αυτό δεν έχει άμεση σχέση με την κυκλοφορία των πολιτών, όμως έχει σχέση με τους πολίτες οι οποίοι κατοικούν και διαμένουν και εργάζονται σε μια χώρα και χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ε, για διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές. Και πάλι εδώ διαγράφεται ένα τεράστιο πρόβλημα. Στην προσπάθεια εισαγωγής κάποιου είδους εναρμόνισης. Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα νομοθετικών εξελίξεων όταν προσπαθείς να συγκεράσεις πολλά, πολλά λεπτομερή προβλήματα ιδίως όσον αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία ε, ε, για το διαδίκτυο η οποία εξελίσσεται συνεχώς ε, και συζητιέται. Από τη μία πλευρά προσπαθούμε να επιτύχουμε πολιτικούς στόχους, δηλαδή να μπορέσουμε να εναρμονίσουμε, κάτι να κάνουμε για την εναρμόνιση του ιδιωτικού δικαίου. Από την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχει και το οικονομικό κίνητρο η ιδέα είναι ότι αν μπορέσεις να εναρμονίσεις ε, τις πτυχές του ιδιωτικού δικαίου θα αυξήσεις τις συναλλαγές, θα αυξήσεις ε, το τζίρο, θα αυξήσεις τα οικονομικά ωφέλη. Και το τρίτο, ο τρίτος στόχος είναι να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των ε, καταναλωτών. Από όλε τι πλευρέ λοιπόν εκφράζονται παρατηρήσει και επικρίσει για αυτού του είδου τι εξελίξει. Ε, προσπαθούμε δηλαδή να καταφέρουμε κάτι μέσω του τετραγωνισμού του κύκλου και να επιτύχουμε διαφορετικούς στόχους ταυτόχρονα. Και το επόμενο θέμα που θέλω να αναφέρω είναι και αυτό το οποίο πιο άμεσα αναφέρεται στη συζήτησή μας μέχρι τώρα, είναι το θέμα της νομολογίας, ε, της ε, πρόσφατης νομολογίας η οποία αναφέρεται στα δικαιώματα εισαγένειας και κυκλοφορίας. Διότι εισαγένεια και δικαιώματα διαμονής είναι μια περίφημη περίπτωση, Σομπράνο, όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε μια πολύ σημαντική απόφαση και αυτή η απόφαση σχολιάστηκε, αναλύθηκε σε πάρα πολλούς ακαδημαϊκούς κύκλους, δεν ήταν όλοι ευτυχείς με την απόφαση, αλλά η ουσία είναι ότι το δικαστήριο έκανε μια πάρα πολύ ισχυρή δήλωση που σημαίνει ότι όταν λέμε ευρωπαϊκή ηθαγένεια, το κεντρικό σημείο της Ιθαγένειας αυτής εστιάζεται στο δικαίωμα διαμονής, δικαίωμα διαμονής και κυκλοφορίας. Αυτό είναι ο πυρήνας της ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Ένα άλλο στοιχείο που έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ζανία που ανέφερε και ο Τόνι είναι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και εκεί θα διαπιστώσετε ότι η συζήτηση μεταξύ ακαδημαϊκών έχει φέρει στην επιφάνεια άλλο ένα πρόβλημα. Είναι το εύρος, το εύρος της εφαρμογής, το εύρος της ε, ισχύω. Σε πολλές ε, περιπτώσεις ήδη έχουμε συζητήσει αν σε αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις εμπλέκονται ευρωπαϊκά δικαιώματα, διότι πολλές φορές οι πολίτες μας δεν ξέρουν πού να στραφούν για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Εάν λοιπόν υπάρχει μια συγκεκριμένη περίπτωση όπου ένας πολίτης έχει περάσει ας πούμε τα σύνορα μεταξύ δύο χωρών ευρωπαϊκών ε, ήδη εμπλέκονται ε, πολλαπλές διαδικασίες. Αλλά στο θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν ξέρουμε εάν μια συγκεκριμένη φράση που χρησιμοποιήθηκε σε σχέση με το ευρωπαϊκό κράτος μέλος είναι η ίδια φράση η οποία έχει ακριβώς την ίδια ισχύ διασυνοριακά ή αλλού. Αυτό ακριβώς εννοώ με την ισχύ, με το εύρος της ισχύω. Πού ισχύει δηλαδή. Ε, καταλαβαίνετε σε τι λεπτομέρεια και σε τι βάθος πρέπει να μπουν οι ακαδημαϊκοί, μια σχολαστικότητα δηλαδή, ε, και αυτός είναι ο τομέας μου και αυτό θα εξετάσω ακριβώς στις μελλοντικές εξέσεις και συζητήσεις. Αυτό το εύρο εφαρμογής, το εύρο ισχύω του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να διευκρινιστεί πλήρως, διότι υπάρχει σχετική ασάφεια. Και τέλος, μια που έχω την ευκαιρία ε, και έχω το λόγο τώρα, αν και μπορεί να επανέλθουμε το απόγευμα, έχει σχέση με αυτό που ανέφερε και ο Τόνι. Τι σημαίνει ηθαγένεια. Έχω κάνει δελεχή έρευνα για, στην ε, συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, στα σημεία που αναφέρεται ακριβώς αυτή η ιδιότητα της ηθαγένεια. Και υπάρχει ασάφεια. Σε πολλά σημεία η ιδιότητα της ηθαγένειας δεν αναφέρεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως εμείς εννοούμε την υπηκότητα ε, που έχει κάποιος ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή με την έννοια των πολιτικών δικαιωμάτων, εάν είμαστε υπήκο ένας κράτος μέλος ή όχι. Γι' αυτό θα ήθελα στις επερχόμενες συζητήσεις να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου θα ενισχύσουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά ενισχύοντας αυτά τα δικαιώματα θα δημιουργήσουμε ε, μία διαμάχη μεταξύ της υπηκότητος και της ηθαγένειας. Διότι μην ξεχνάτε ότι υπάρχει το καυτό θέμα των επικών τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια ως ξένοι ως αλλοδαπή πάρα πολλά χρόνια και θέλουμε σε πολλές περιπτώσεις να τους βοηθήσουμε μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της ε, ευρωπαϊκής ιδιότητας, της ιδιότητας δηλαδή του κατοίκου, αν, όχι, αν και όχι ε, ηθαγενούς ή ε, υπηκόου το, το, λεπτό ζήτημα είναι ε, κάποιος ο οποίος διαμένει μακροχρόνια στην επικράτειά μας πρέπει να τύχει της ίδιας μεταχείρισης όπως ένας Ευρωπαίος Ιθαγενής που έχει την Ιθαγένεια. Πολλές φορές λοιπόν δεν γίνεται η μεταχείριση, υπάρχει μεγάλη διάκριση παραδείγματο χάρη στο, ένταλμα, στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης όπου ένας Ιταλός υπήκος Α, όπου ένας αλλοδαπός τρίτης χώρας είχε διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα, τέτοιου βάρους δηλαδή στην Ιταλία που το Ιταλικό Δικαστήριο ε, ότι μπορεί και πρέπει να απελαθεί διότι δεν την χάνει, δεν καλύπτεται από τα δικαιώματα της, ε, του Ευρωπαϊκού ε, του Ευρωπαίου πολίτη και του θεμελιώδους χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, εκεί λοιπόν βλέπετε τι διαφορές προκύπτουν. Και το δικό μου επιχείρημα λέει ότι δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή οικοδομούμε κάτι, ίσως τα επόμενα χρόνια, πέντε χρόνια, δέκα χρόνια, να εδρεωθεί επιτέλους η ευρωπαϊκή ε, ηθαγένεια πέραν των κρατών, μελών και πέραν της έννοιας της στενής εθνικότητας. Αυτά είχα να πω κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε βέβαιος ότι το πανεπιστημιακό βλέμμα έχει τη θέση του στη συζήτηση αυτή. Υπάρχει αυτή η εναρμόνιση βεβαίως, αλλά είναι τόσο περίπλοκη να την επιτύχουμε με όλες αυτές τις ε, διάφορες νομοθεσίες ε, που πρέπει να τις ε, συγκεράσουμε. Το πρόβλημα της επικουρικότητας που, που και που το αναφέρουμε είναι ένα σημαντικό φρένο της εφαρμογής του, της νομοθεσίας που αφορά τον πολίτη νομίζω ότι θα είναι αντικείμενο τη συζήτηση και χάρηκα ιδιαίτερα που αναφερθήκατε στο θέμα της, ε, του εντάλματο συλλήψεω, ε, γιατί πραγματικά μερικές φορές γίνεται κατάχρηση για προβλήματα ποινική φύσεως συνήθως ε, και χρησιμοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όμω, ενδεχομένως να επανέλθουμε και σε αυτό στη συζήτηση. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον τελευταίο μα ομιλητή, τον Πολ Νέμιτς, ο οποίο είναι διευθύντη ε, θεμελιώδη δικαιώματα και ηθαγένεια τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κύριε Νεμίτ, ε, ε, θα ήθελα να σα δώσω το λόγο για πέντε λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το ευρωπαϊκό έτος του πολίτη σήμαινε διαβούλευση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και το Κοινοβούλιο γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί σας σήμερα σε αυτήν την αποκοινού ε, σε αυτή την κοινή ακρόαση το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας πω ορισμένα πράγματα τα οποία είπε και η Φρονσουάζ Λεμπά είπε στην αρχή και άλλωστε θα τα πει και στο τέλος ε, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, η κυρία Ρέντινγκ. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία δεν έχουν ακόμη αναφερθεί. Πρώτον, όταν πρόκειται για την επιβολή του ευρωπαϊκού, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, που, κάτι που δεν αναφέρθηκε και κάνει και τη, είναι και η διαφορά μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, οποιασδήποτε άλλη συνεργασίας μεταξύ κρατών, περιφερειών κλπ. είναι ότι ο εθνικός δικαστής είναι αυτός που ερμηνεύει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο εθνικός δικαστής πρέπει να παρέχει αυτά τα δικαιώματα που ε, υπόσχεται το ευρωπαϊκό δίκαιο στον πολίτη. Ναι, θέλουμε να μιλάμε για τις δικές μας δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής Αναφορών του Κοινοβουλίου κλπ. Όμως, ο μοναδικός παίκτη στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που μπορεί να παρέχει το δικαίωμα σε έναν πολίτη με απόφαση είναι ο Εθνικός Δικαστής. Γιατί ακόμη και αν η Επιτροπή αρχίσει μια διαδικασία επί παραβάση και ακόμη και αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι ορθώς το έκανε αυτό ε, το κράτος, ότι ορθώς το έκανε το κράτος, ε, ο εθνικός δικαστής είναι αυτός ο οποίος μπορεί να διατάξει το κράτος ε, να υποχρεώσει το να, να παραχωρήσει το δικαίωμα αυτό, όμως δεν μπορεί να το κάνει απευθείας στον πολίτη. Δεν μπορεί να πει δηλαδή εφαρμόστε αυτό το δικαίωμα, αλλιώς θα έρθει ο δικαστικός κλητήρας να σας πάρει. Οπότε πρέπει να το υπενθυμίσουμε αυτό το σημαντικό στοιχείο ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ άλλων μορφών ε, ολοκλήρωσης και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι ότι στις άλλες ότι, ότι, ότι ε, είναι απευθείας ε, εφαρμοστέο και μπορεί ο πολίτης να πάει στον Εθνικό Δικαστή να ζητήσει κάτι τέτοιο. Όταν μιλάμε λοιπόν για την επιβολή του νόμου είναι σημαντικό αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώνουμε τις εθνικές ε, ε, κυβερνήσεις, η επικουρικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικά, σημαντική, είναι πράγματα στα οποία επενδύουμε βεβαίως, αλλά να μην ξεχνούμε ότι η δραστηριότητα της εθνικής ε, διοίκηση ελέγχεται από τον Εθνικό Δικαστή και έχουμε πάρα πολλές αποφάσεις που έχουν ε, ληφθεί κατόπιν προδικαστικού ε, αιτήματο στο πλαίσιο του δικαστηρίου σε σχέση με την επιβολή του νόμου από τους εθνικούς δικαστές. Δεύτερον, είναι σημαντικό τα δικαιώματα ηθαγένειας ε, ε, πρέπει να είναι ελκυστικά και για όσους δεν, τους δεν τα χρησιμοποιούν. Και τι εννοώ με αυτό. Αυτό που εννοώ είναι ότι όταν έχουμε 500 εκατομμύρια κατοίκου, έχουμε, τουλάχιστον, έχουμε λιγότερους από 20% που χρησιμοποιούν αυτά τα δικαιώματα που έχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μονίμως. Αυτό όμω είναι μια μικρή ομάδα μέσα στα 500 εκατομμύρια και γι' αυτό πρέπει να εξηγήσουμε, να επιχειρηματολογήσουμε γιατί οι άνθρωποι που είναι σπίτι του έχουν συμφέρον να δουλεύει κάτι τέτοιο. Και αυτά νομίζω τα επιχειρήματα έχουν όντω παρατηθεί. Πρέπει όμως να τα φέρουμε στο προσκήνιο. Γιατί? Γιατί σε περίοδο οικονομική κρίσης χρειαζόμαστε την κινητικότητα των ανθρώπων που θα αντισταθμίσει το γεγονός ότι σε αντιπαραβολή με άλλε υπήρου μειώνεται ο πληθυσμός ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό σημαίνει μείωση της ανάπτυξης και αυτό σημαίνει μείωση των θέσεων απασχόλησης και αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί, αντισταθμιστεί μόνο με την κινητικότητα, την έρευνα, την καινοτομία και γι' αυτό ακριβώς πρέπει αυτό το επιχείρημα να το περάσουμε σε όσους είναι στο σπίτι τους και πρέπει να το κάνουμε στην πράξη. Αυτή είναι ε, η άποψή μου και, θα ήθελα να σας το πω και να την ε, εξηγήσω και σε εσά. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να υποδεχθούν τους ανθρώπους από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και αυτοί οι οποίοι είναι οι πιο ευχάριστοι, οι πιο ανοιχτοί. Σκεφτείτε το Αμβούργο, σκεφτείτε το Λονδίνο. Ε, το Αμπουσταμβούργο αποφάσισε ο Δήμαρχος ε, σε όποιον θέλει να δώσει ε, ηθαγένεια εάν βέβαια το επιτρέπει και η νομοθεσία της χώρας προέλευσής του. Λοιπόν πρέπει να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, να δείξουμε ότι αυτά τα δικαιώματα, τα δικαιώματα ηθαγένειας, ελεύθερης μετακίνησης είναι καλά ακόμη και για τους ανθρώπους που δεν τα χρησιμοποιούν. Γιατί αυτή είναι η μεγάλη πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά είναι τα οικονομικά επιχειρήματα, αλλά πρέπει να έχουμε και επιχειρήματα μιας ανθούσας κοινωνίας. Είναι πάρα πολύ καλή η κινητικότητα για όλους, για την ποιότητα της ζωής και είναι και διασκεδαστικό για να το πω και απλά. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να αξιολογήσουμε και να κάνουμε αυτή τη σύνδεση μεταξύ του πολιτισμού υποδοχής στις πόλεις και στις χώρες και από την άλλη την οικονομική ε, απόδοσή τους και την ε, απόδοσή τους ε, στην καθημερινή του ζωή. Πρέπει να δούμε και τις διάφορες μεθοδολογίες για το πώς μπορούμε να εξετάσουμε το θέμα αυτό. Άκουσα πολλές καλές ιδέες εδώ σήμερα και νομίζω ότι θα έπρεπε στο ε, πλαίσιο της επικουρικότητας πρέπει σε διάφορες περιφέρειες να δοκιμάσουμε διάφορους τρόπους οργάνωσης της αυτοδιοίκησης, της ενημέρωσης κλπ. Και από καιρού εις καιρών πρέπει να τις αντιπαραβάλουμε, να δούμε τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει. Νομίζω ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να προσπαθήσουμε να όλες όλες αυτές τις διαδικασίες ε, ε, εισαγωγής στα διάφορα επίπεδα ε, της διοίκησης να τις ρυθμίσουμε από τις Βρυξέλλες με διάφορους τρόπους. Ακούσαμε από τον κύριο Παράτη ένα παράδειγμα 72 ε, ώρες στην ε, Ολλανδία, πολύ περισσότερο στο Βέλγιο μπορεί να πάρει αυτή η διαδικασία. Και πρέπει όλα αυτά τα ζητήματα να τα λάβουμε υπόψη, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ιδιαιτερότητες. Το είπατε και εσείς κύριε Κάσουμαν, είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι ιδιαιτερότητες. Παράλληλα όμως πρέπει να σκεφτούμε και τον κανόνα των μεγάλων αριθμών, αλλά και τις βασικές αρχές. Η άποψή μου λοιπόν θα ήταν σε αυτό το τεράστιο θέμα της ηθαγένειας πρέπει να κάνουμε και τα δύο. Σε αυτή τη συζήτηση για την ηθαγένεια πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες αλλά πρέπει να σκεφτούμε και ποια είναι τα, θέματα που αφορούν την πλειοψηφία των πολιτών και ποιες είναι οι βασικές αρχές. Και λειτουργούν αυτές οι αρχές. Και θα έλεγα ότι σε αυτό το σημείο δεν τα πάμε και τόσο άσχημα. Άκουσα πάρα πολύ συγκεκριμένα σημεία από το πάνελ και βεβαίως ε, δεν μπορώ να σας διαβάσω διεξοδικά την, ε, την, ε, τον κατάλογο της έκθεσης Περιθαγένειας του 2010 ε, 10, συγγνώμη, και αυτά που μας είπε η κυρία ε, Κοράτσα Μπίλτ. Ε, ε, φυσικά θα μπορούσα να αναφερθώ στις ε, πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το, τους ομοφιλόφιλους, το διάλογο που είχαμε με την Ισπανία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτό αυτό τον κανόνα των βασικών αρχών αλλά και των μεγάλων αριθμών στο μυαλό μας. Γιατί μερικές φορές υπάρχει ένας πειρασμός ε, αυτές τις βασικές αρχές να τις αμφισβητήσουμε ευρύτατα και θα ήθελα με αυτό να ολοκληρώσω. Όταν λοιπόν τίθενται να αμφιβόλω οι βασικές αρχές, χρειαζόμαστε δέσμευση, όχι μόνο μέσω ψήφου, αλλά χρειαζόμαστε νέες ιδέες, πώς μπορούμε να ε, προχωρήσουμε, αλλά πώς μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε και όλα αυτά τα οποία έχουμε ήδη επιτύχει. Γιατί α μην γελιόμαστε, η οδηγία για την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι τεράστιο επίτευγμα, πολύ ε, βιώσιμη σε πολλέ χώρε μέλη. Εντάξει, πρέπει να συζητήσουμε βέβαια για ε, το πώ θα είναι η επόμενη συνθήκη και ναι, όντω θα γίνει ε, μία πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλο του 2013, αρχέ του 2014, Όμω, δεν πρέπει μόνο να ασχοληθούμε με τα θέματα τη οικονομική διακυβέρνηση, που είναι βέβαια ένα τεράστιο κομμάτι τη όλη διαδικασία αλλά πρέπει από την άλλη να αντιμετωπίσουμε και ορισμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των πολιτών. Παράλληλα όμως, ότι αυτά που έχουμε ήδη στην οδηγία αξίζει τον κόπο να τα διατηρήσουμε. Τελειώνω λοιπόν λέγοντας για, τα κοινωνικά μίντια και, και τη δημοκρατία. Έχουμε το hashtag στο Twitter EYC e 2013. Ε, αυτό είναι το hashtag μας στο, στο Twitter. Παρακαλώ να συμμετέχετε στη συζήτηση και εκεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νέμιτς για τα όσα μας είπατε. Θα ξεκινήσει τώρα η συζήτηση μεταξύ ημών. Μη διστάσετε να λάβετε το λόγο, να μας πείτε τις ιδέες σας, τις μαρτύριες σας, τις προτάσεις σας, τα βιώματά σας, τα ερωτήματά σας. Μη διστάσετε να θέσετε ερωτήματα στους ομιλητές μας. Αν έχετε μια ερώτηση για κάποιον συγκεκριμένα, ε, παρακαλώ να μας το πείτε όταν θα λάβετε το λόγο. Ήθελα να δώσω το λόγο, καταρχάς, στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά κάποιοι απουσιάζουν. Ε, κάποιοι άλλοι ελπίζω να έρθουν εντωμεταξύ, αλλιώς ε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα ήθελα, όποιο λάβει το λόγο, σα παρακαλώ να μιλάει για δύο λεπτά το πολύ. Μπορείτε να μιλήσετε λιγότερο, αλλά όχι πάνω από δύο λεπτά. Για να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερε ε, ε ομιλίε. Έχουμε και ένα σχόλιο από την Μπέρμπαρα Σνάιντερ στο Twitter. Θα το αναφέρω, αν θέλει κάποιος να ε, απαντήσει και αλλιώς ε, θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Σίλων. Η Γερμανία, παρά το γεγονός ότι απογράφει τα πρωτόκολλα 7 και 12 για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την οικογένεια και τις διακρίσεις, δεν τα έχει ακόμα κυρώσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δράσει για να συμπληρωθεί αυτό το κενό. Η Κομισιόν, μήπως θέλει να απαντήσει θα πρέπει να το εξετάσω κατά πόσον υπάρχει υποχρέωση μέσω Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για κύρωση αυτών των συμβάσεων. Κύριε Σόγκορ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Δεν έχω ερώτηση. Απλώς ε, θα ήθελα να πω κάτι σε συνέχεια της παρέμβασης του κυρίου Νέμιτς. Ήμουν 7 χρόνια γερουσιαστή στην ε, χώρα μου και δεν μπορούσα να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Θα τη χρησιμοποιήσω λοιπόν τώρα και θα μιλήσω ουγγρικά. Ο κύριος Νέμιτς αναφέρθηκε σε κάτι σημαντικό. Οι πολίτες οι οποίοι δεν επιθυμούν να φύγουν από τη χώρα τους, που δεν θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, αλλά δεν μπορούν και να ασκήσουν το δικαίωμα της χρήσης της μητρικής τους γλώσσας. Είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας γιατί είναι αντικείμενο διακρίσεων στο χώρο της εργασίας τους, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, την ε, εθνική τους γλώσσα. Εγώ είμαι από την Ανατολική Ευρώπη και στη χώρα μου δεν έχω με αυτό το πρόβλημα, αλλά υπάρχουν πολίτες οι οποίοι είχαν ιδιοκτησία στη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος και δεν μπόρεσαν να ανακτήσουν την ιδιοκτησία τους. Την έχασαν και τώρα δεν μπορούν να την ανακτήσουν. Πρόκειται λοιπόν για πολίτες που έγιναν πολίτες άλλης χώρας και αναφέρομαι και σε αυτά τα δικαιώματα. Πρόκειται για μειονότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει ε, προφανώς να ενθαρρύνουμε τους πολίτες μας να ζουν με ευρωπαϊκό τρόπο και εγώ ως ε, σκιώδης εισηγητής ε, και θα σταθεί και αυτό η συνάδελφός μου σήμερα το απόγευμα διότι έχουμε το ευρωπαϊκό έτος Ευρωπαϊκή Υπηκότητα. Εγώ ήμουν ασκιώδη εισηγητή και είχα πολλέ δυσκολίε, διότι δεν μπορώ να πω στου πολίτε μα που βρίσκονται στις χώρες τους, γιατί γίνεται συνεχώς διάκριση. Εμείς γεννηθήκαμε εκεί, στη χώρα μας και θέλουμε να παραμείνουμε στη χώρα μας. Πρόκειται λοιπόν για εθνικές μειονότητες, είμαστε μια μειονότητα περίπου 7% και ε, νομίζω ότι για παράδειγμα στην Ιταλία λιώθηκε με πολύ καλό τρόπο το θέμα των μειονοτήτων. Θα πρέπει να γίνει κάτι και στις άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Κύριε Νέμιτς, ε, σας ευχαριστώ πολύ για την ε, ερω... παρέμβασή σας. Είναι όντως πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περιορίζει την ελευθερία των κρατών μελών να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που απαγορεύουν τις διακρίσεις υπάρχουν κανόνες που επιβάλλουν ε, την ελευθερία κυκλοφορίας ακόμα και σε ομόφυλα ζευγάρια και σε άτομα τα οποία έχουν σύμφωνο συμβίωσης. Αυτό είναι ελευθερία. Δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διάκρισης. Αυτό που περιγράφετε εσείς είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε, θα μπορούσε ε, επαναλαμβάνω, να αναφέρεται στο άρθρο 7 της ε, ε, συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί το αποκαλούν ατομική βόμβα αυτό το άρθρο, αλλά καταδεικνύει ότι υπάρχουν και περιορισμοί προς τα κράτη-μέλη που σχετίζονται με βασικές αρχές διακρίσεων, δημοκρατίας και ούτω και νομίζω ότι στη διάρκεια του τελευταίου 1,5 χρόνου, δηλαδή από τότε που τέθηκε σε η δεσμευτική χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέδειξε ότι ακολουθούμε αυτή τη νέα κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μία οικονομική και μόνο ένωση, αλλά μία ένωση βασικών αρχών και θεμελιωδών δικαιωμάτων και αυτό το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Και εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε λάβει μέτρα για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία. Ε, υπάρχουν ακόμα και δικαστικές διαδικασίες στην Ουγγαρία, όταν υπήρχε φυσικά νομική βάση προς αυτό. Ε, θα πρέπει να είναι σαφές βέβαια ότι ε, έχουμε κάποιες περιπτώσεις τις οποίες δεν υπάρχει νομική βάση και εκεί δεν μπορούμε να δράσουμε νομικώς. Και αυτή είναι και η συνήθις αρχή περιορισμού της εξουσίας. Η εξουσία θα πρέπει να εγγράφεται στο δίκαιο. Ευχαριστώ κυρία Νέμιτ και κυρία Βαλεάν θέλει να απαντήσει. Actually something to respond to. Θα ήθελα και εγώ να απαντήσω σε κάτι γιατί αυτή είναι μια περίπτωση την οποία όλοι γνωρίζουμε. Υπάρχουν μειονότητες, υπάρχουν τα εθνικά κράτη-μέλη που έκανε ένα δημοψήφισμα πρόσφατα στην Καταλωνία. Στη Σκοτία προτείνεται κάτι τέτοιο. Αυτό δείχνει ότι προκύπτουν διάφορα ζητήματα προς συζήτηση, το Ηνωμένο Βασίλειο, αν η Σκωτία είναι μέρος, δεν είναι κλπ. Αυτά όλα συνάδουν με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη έχουν οργανωθεί. Κατηδίαν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κράτος μέλος ε, κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μόνο ένα, ας πούμε, ή ένα συγκεκριμένο κάνει αρνητικές διακρίσεις ε, κατά το, των πολιτών του. Ε, δεν είναι λοιπόν ε, ένα θέμα το οποίο επιβαρύνει ένα κράτος μέλος μόνο. Είναι ένα θέμα γενικό το οποίο δείχνει ότι υπάρχουν μειονεκτήματα στον τρόπο διοργάνωσης ενός κράτους. Υπάρχουν ε, μια οργάνωση, μια υποδομή ενός κράτους μπορεί να επικεντρώνεται στη περιφερειακή διοίκηση, μπορεί να είναι αποκεντρωμένη, ε, μπορεί να δίνει ιδιαίτερη σημασία στο δικαίωμα εκπροσώπησης, παραδείγματο χάρη στις μειονότητες στην Ουγγαρία, όπως είπε και ο συμπατριώτης μου, ήταν γερουσιαστής για πολλά χρόνια και δεν μπορούσε να μιλήσει τη γλώσσα του, αυτή τη στιγμή τα τελευταία 15-20 χρόνια η ουγγρική μειονότητα εκπροσωπείται στο ουγγρικό κοινοβούλιο. Πάντοτε βεβαίως θα υπάρχει παράπονο, πάντοτε θα υπάρχει κάτι που σηκώνει βελτίωση. Αυτό μπορεί να συζητηθεί στα εθνικά κοινοβούλια. Το Εθνικό Κοινοβούλιο μπορεί να συζητήσει και να αποφασίσει εάν θα παράσχει το ένα ή το άλλο δικαίωμα. Άρα λοιπόν λοιπόν δεν πρέπει να συζητήσουμε ε, ξεχωριστά για τους, ε, τις ευρωπαϊκές μειονότητες. Ε, τα δικαιώματα των μειονοτήτων καλύπτονται από τους καταστατικούς χάρτης και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε κάθε κράτος μέλος. Εάν λοιπόν λάβουμε ε, υπόψη τα, τους, τα μεγάλα αριθμητικά στοιχεία, ε, θα χάσουμε ίσως από τα μάτια μας ε, τις, τις μικρές ομάδες. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε με μικρά ή μεγάλα νούμερα, αλλά με προσωπικές περιπτώσεις. Εγώ αυτό υποστηρίζω. Εάν ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πρόβλημα ως προς την, το σεβασμό των δικαιωμάτων του, πρέπει να χειριστούμε αυτή την υπόθεση του μεμονωμένου πολίτη και όχι του πολίτη αυτού ως μέλους μιας άλλης ομάδας, μιας άλλης κοινότητας ή μιας μειονότητας. Κατά περίπτωση λοιπόν ως Ευρωπαίου πολίτη πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα παράπονά του και τις προσφυγές του και τα δικαιώματά του όταν καταγγέλλονται. Ευχαριστώ πολύ. Η, διαφορά είναι ότι με μία αναφορά μπορεί κάποιος ε, ε, πολίτης να ζητήσει ε, τοποθέτηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι διαφορετικό βέβαια από την κοινωνία, από την πρωτοβουλία των πολιτών. Κύριε Κάσμαν, ευχαριστώ. κύριος Κάσμαν. Και εγώ απηχώ εν μέρει αυτά, τα, ασπάζουμε μάλλον εν μέρει αυτά τα οποία και η Ρία Βάλεαν. Ε, αυτά τα θέματα καλύπτονται από τις αρμοδιότητες ε, των κρατών μελών. Σε αυτές τις αρμοδιότητες νομικά δεν μπορεί να παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο χάρτης των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων εφαρμόζεται μόνο στο πεδίο εκείνο στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα. Παραδείγματο χάρη, δεν μπορεί να παρέμβει μεμονωμένα σε εργασιακά θέματα στον τόπο εργασία. Αυτό όμως είναι ακριβώς ένα μέρος του προβλήματος. Όταν αποφασίσαμε τη διεύρυνση, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μισό εκατομμύριο απάτριδες οι οποίοι είναι, ε, κατοικούν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν μπορούν να μετακινηθούν, δεν έχουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, δεν έχουν τα δικαιώματα που πρέπει να έχουν. Έχουμε αποτανθεί στην Κομισιόν, η Κομισιόν το γνωρίζει, τα θεμελιώδη όργανα το γνωρίζουν, αλλά δεν έχουν κάνει τίποτα γι' αυτό. 500.000 άνθρωποι στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν καν την ιδιότητα ε, τη ηθαγένεση του Ευρωπαίου πολίτη. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να προβάλλουμε στην πλειοψηφία των πολιτών μας ε, τα πλεονεκτήματα και τα ωφέλη που προκύπτουν από μία ενσωματωμένη, ολοκληρωμένη και εις βάθος εφαρμογή ε, της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας διότι στο τέλος της ημέρας οι δημοκρατίες κρίνονται από το πώς χειρίζονται όχι τις πλειοψηφίες αλλά τις μειοψηφίες, τις μειονότητες. Άρα λοιπόν τα ωφέλη της ενσωμάτωσης και της συμπερίληψης όλων είναι τεράστια. Πρέπει όμως να προβάλλονται και ε, να δίνεται η μάχη για την προάσπισή τους από θαραλέους ε, πολιτικούς είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε πολίτες οι οποίοι υποβάλλουν τις αναφορές τους και έρχονται σε επαφή άμεσα με μας, ώστε οι αναφέροντες να μπορούν να μας εξηγήσουν κάτι διάν, τι συμβαίνει ε, και πώς θίγονται ή παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. Και θα ήθελα να σας ζητήσω να πάρτε όλοι αυτή την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών για να δείτε ακριβώς πώς, τι, τι ωφέλη προκύπτουν από την ενεργό εφαρμογή των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Ο πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση αυτή. Μήπως θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος να πάρει το λόγο. Θα ήθελα τότε για τρία λεπτά να πω ότι δεν υπάρχει μόνο η ελευθερία της κυκλοφορίας ε, που δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχει επίσης και η προστασία του άμεσου περιβάλλοντος του Ευρωπαίου πολίτη και η μεγαλύτερη, ε, η πληθώρα των αναφορών στην Επιτροπή Αναφορών αφορούν ε, τα, το περιβάλλον ε, και τα προβλήματα κυκλοφορίας. Όντως, Βλέπουμε ας πούμε την μη, το μη σεβασμό της οδηγίας Natura 2000 ε, για το, τα οικοσυστήματα κλπ που δεν εφαρμόζονται ε, στα κράτη-μέλη ε, και αυτό εμφανίζεται συνεχώς, επανέρχεται συνεχώς στην Επιτροπή Αναφορών. Συνήθεις απαντήσεις που δίνουμε στους αναφέροντες είναι ότι πρέπει πριν έρθουν σε εμά να εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες προσφυγής ε, στο πλαίσιο της χώρας τους. Και για έναν Ευρωπαίο πολίτη αυτό είναι πολύ ε, μακρόχρονη διαδικασία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει επικουρικότητα, το εθνικό δίκαιο, το συζητήσαμε και προηγουμένως, αλλά μήπως θα μπορούσαμε να προβληματιστούμε εδώ από κοινού, να δούμε πώς μπορούμε να επισπεύσουμε λίγο αυτές τις ε, διαδικασίες ε, στην Επιτροπή Αναφορών. Πολλοί αναφέροντες, ε, όπως είπε και ο Μάικλ, έρχονται να μας συναντήσουν απευθείας και στους οποίους λέμε και εκεί τους απογοητεύουμε γιατί υποχρεωνόμαστε να τους πούμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής θα Ιθαγένους απογοητεύουμε για να τους πούμε είναι πάρα πολύ νωρί να έρθείτε σε εμά. κάντε όλες τις διαδικασίες στη χώρα σας και μετά θα έρθείτε σε εμά για να ε, μας ρωτήσετε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ρωτώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένοντας την απάντησή της είναι πραγματικά μια διαδικασία πολύ ε, σημαντική. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν προβλήματα περιβαλλοντικά τεράστια που αναφέρονται στην Επιτροπή Αναφορών και το δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι βέβαια στην προάσπιση του δικαιώματος ε, του Ευρωπαίου πολίτη ο συνήγορος του πολίτη σε κάθε χώρα είναι ένα ε, πρόσωπο πάρα πολύ σημαντικό και εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ με τους συνήγορους του πολίτη και με τον Ευρωπαίο Διαμισολαβητή ε, από κοινού ε, στο πλαίσιο της ε, Επιτροπής Αναφορών, ε, η οποία κάνει έτσι μια δουλειά εξαιρετική. Κρίμα που δεν υπάρχει συνήγορος του πολίτη σε, όλους, σε όλα τα κράτη-μέλη. Εμείς έχουμε κραυγαλαίες περιπτώσεις. Ε, ε, μιλάω για το Jugendamt για παράδειγμα, ένα πρόβλημα διακρατικού διαζυγίου που αφορά κυρίως την ε, ε, Γερμανία. Αρχίζουμε να έχουμε και κάποιες περιπτώσεις στη Δανία, αλλά βασικά αφορά την Γερμανία. Υπάρχουν κατάφορες παραβιάσεις δικαιωμάτων οι οποίες θα μπορούσαν να επιληθούν από τον συνήγορο του πολίτη στη Γερμανία. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σε δύο από τις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μου φαίνεται στην εποχή μας εντελώς ε, τεράστια δυναμία, τεράστιο κενό, ειδικότερα όταν θέλουμε να προοδεύσουμε με την ευρωπαϊκή Ιθαγένεια δεν είναι τόσο ερώτημα, είναι περισσότερο παρατήρηση των όσων έχουμε ζήσει ε, και στο πλαίσιο της Επιτροπής των Αναφορών και αν κανείς δεν θέλει να πάρει το λόγο, θα ήθελα να δώσω το λόγο σε οποιονδήποτε από την αίθουσα θέλει να ε, μιλήσει, όχι πάνω όμως από δύο λεπτά. Η Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή. Είμαι πρόεδρος της Οικονομικής Κίνησης και μέλος της ε, Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Ε, okay. Θα ήθελα να αναφέρω δύο επιτυχή παραδείγματα για να ε, δημιουργήσουμε πραγματικά ένα επιτυχημένο κράτος για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Το πρώτο το πρώτο που πρέπει να πω είναι ότι υπάρχει μία έχει διαμορφωθεί μία ε, αντίληψη ενεργούς ε, συμμετοχής, ενεργούς ηθαγένειας, ε, δραστηριότητας και δεν πρέπει να τονίζουμε μόνο τα αρνητικά εμπόδια, τις αρνητικές πτυχές. Λοιπόν, πώς θα επιτύχουμε. Πρώτον, βεβαίως, με το να απαλείψουμε κάθε έννοια πολιτών δεύτερης κατηγορίας Ξέρουμε ακόμα ότι στην Κύπρο δεν μπορεί να μετακινούνται, να κυκλοφορούν οι πολίτες ελεύθερα μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Και στη Λετωνία ξέρω ότι υπάρχουν άτομα τα οποία παίρνουν τις μισές επιδοτήσεις από ότι άλλοι αγρότες ή παραγωγοί, αλλά πρέπει να ανταγωνιστούν στις ίδιες αγορές. Άρα λοιπόν πρέπει και αυτοί να έχουν το δικαίωμα να είναι ανταγωνιστική. Η κοινωνία των ε, πολιτών, ε, χρηματοδότηση. Όσοι είναι εδώ στην αίθουσα πρέπει να ξέρουν. Εμείς είμαστε οι συνήθεις ύποπτοι ε, ή είναι οι πολίτες μας σε κάθε χώρα. Όσον αφορά, επαναλαμβάνω, τη χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο εθνικό επίπεδο είναι ένα σημείο κλειδί το οποίο ε, πρέπει να λειτουργεί ομαλά. Το δεύτερο στοιχείο που μπορούμε να ε, βελτιώσουμε είναι η απάλληψη οργανισμών ή φορέων που θεωρούνται ως ε, δεύτερης κατηγορίας, υποδέστερη. Παραδείγματο χάρη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακούγεται και ακούει, ακούει τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό εδώ που γίνεται σήμερα είναι μία σημαντική πρωτοβουλία για να ακουστεί και η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών και οι επικρίσεις που έχουν στο σώμα. Δύο προτάσεις συνεργασίας. Πρώτον, η συμμετοχική δημοκρατία και ενεργό συμμετοχή. Θα πρέπει να υπάρχει μία ε, προσέγγιση τύπου αγοράς ε, στο οποίο ε, να μπορεί να γίνεται ακριβώς αυτή η κοινή συζήτηση μεταξύ των φορέων ε, και των πολιτών. Αγορά, αγκόρα. Και ότι αυτή η διοργάνωση θα παίξει ένα μεγαλύτερο ρόλο. Αυτή τη στιγμή 56 ε, οργανισμοί και φορείς συμμετέχουν σε αυτή την ευρωπαϊκή αγορά, ε, το, το φόρουμ δηλαδή. Και μπορούμε να ε, βελτιώσουμε τις δραστηριότητες του και την προβολή του. Η άλλη πτυχή είναι η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Παραδείγματο χάρη η πράσινη βίβλος ε, μπορεί να ε, ε, επιτύχει στην εφαρμογή της μόνο εάν όλα τα θεμελιώδη όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργαστούν καλύτερα υπό το πρίσμα του άρθρου 11. Πολλά πράγματα ακόμα συνεχίζουν να γίνονται ή να συζητώνται πίσω από κλειστές πόρτες, ιδίως στο Συμβούλιο, στο Συμβούλιο αλλά και σε άλλους οργανισμούς και σε άλλους φορείς πολλά πράγματα παραμένουν κρυφά κάτω από το τραπέζι. Όλα αυτά πρέπει να βγουν στην επιφάνεια και να βελτιωθεί η επικοινωνία για να ακούγεται η φωνή όλων. Αυτό θα βοηθήσει στην επιτυχία του έτους. Ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις σας και την παρέμβασή σας. Πράγματι, το Κοινοβούλιο στα πλαίσια της συζήτησης για τις πολιτές δημοσιογνωμικές προοπτικές λαμβάνει αυτό υπόψη τους και αυτό δείχνει ότι και στο επίπεδο της συζήτησης για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Εμείς είμαστε πιο ε, ε, φιλόδοξοι στον προπολογισμό, επιστημούσαμε περισσότερη Ευρώπη από ό,τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο στη συζήτηση στους επόμενους μήνες, ε, τι θέλουν οι μεν, τι θέλουν οι δε και ένα, θα είναι ένα τμήμα της ε, στάσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Κορατσαμπίλτε. Φίλιπ, ε, πρέπει να πω ότι έμαθα πολλά και συμφωνάω με τα περισσότερα πώς ακούστηκαν. Καταρχάς, δύο πράγματα. Νομίζω ότι ως νομοθέτες ε, δεν είμαστε βέβαια κατά των ε, διακρίσεων σε καμία περίπτωση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε οι πρώτοι που υψώνουμε τη φωνή μας κατά των διακρίσεων ε, δικαιώματα μειονοτήτων, ζευγαριών ιδίου φύλου και δικαιώματα για όλους, όχι μόνο για τους πολίτες που απλώς κυκλοφορούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτή την άποψη. Επίσης, πρέπει να πω ότι σήμερα φεύγω με μια βαριά ευθύνη για να απαντήσουμε σε περιπτώσεις της δικές, σαν τη δική σας. Να έχουμε πιο οργανισμένα θέματα, να μην έχουμε κατακαιρματισμό και να μειώσουμε την γραφειοκρατία για τους πολίτες. Να μην πρέπει να δίνουν ολόκληρο αγώνα για να αποκτήσουν κάτι δεδομένο. Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υπενθύμησε ότι υπάρχει ένας κατάλογος δράσεων, ένα εξελίξη που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και σίγουρα θα βελτιώσουν τις δυνατότητες των πολιτών η μπλε κάρτα για παράδειγμα, η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ε, και το EMI. Θα ήθελα να ρωτήσω εδώ ε, ποιοι ξέρουν τι είναι το IMI, το Εσωτερικό Σύστημα ε, Πληροφοριών Αγοριών. Αυτό θα αλλάξει τη ζωή σα, το εγκρίναμε, είναι νομοθεσία, εγώ ήμουν σκιώδη εισηγήτρια. Ε, ήμασταν πολύ απογοητευμένοι, πρόκειται για μια νομοθεσία η οποία δεν είναι καθόλου δημοφιλή, αλλά θα αλλάξει τη ζωή των πολιτών. Πώς θα το ε, προωθήσουμε αυτό. Και νομίζω ότι αντί για χάρτα, θα εξετάσω βέβαια την πρότασή σας πολύ προσεκτικά, Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να προβάλλουμε αυτά τα οποία κάνουμε, τι έχουμε επιτύχει και να νιώσουν οι πολίτες ότι υπάρχουν ωφέλη, διότι όλη αυτή η συζήτηση για την ηθαγένεια, αν ε, μιλήσετε με Σουηδούς, οι περισσότεροι Σουηδοί δεν θέλουν να είναι Ευρωπαίοι, θέλουν να είναι Σουηδοί που έχουν δικαιώματα. Και νομίζω ότι ότι αν δεν κατανοήσουμε και δεν δεχθούμε την πρόκληση ότι οτιδήποτε ευρωπαϊκό μπορεί να θεωρείται πρόκληση ή και απειλή για τους πολίτες. Απειλή στη σουηδική τους ταυτότητα ή στην εθνική του ταυτότητα, ε, τον πολιτισμό, την παράδοσή τους. Αν δεν μπορέσουμε λοιπόν εμείς να τους πούμε ότι ενωμένοι στη διαφορετικότητα και διαφορετικότητα σημαίνει ότι σεβόμαστε τους πολιτισμούς και τις παραδόσεις, ε, δεν θα επιτύχουμε. Μπορεί να λέμε εμείς συνέχεια, αλλά ο κόσμος αδιαφορεί. Ε, μπορεί, θα πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε με την εθνική ταυτότητα, τις παραδόσεις, ε, τον πολιτισμό, ακόμα και τις συνταγές και τον τρόπο ένδυσης. Οτιδήποτε είναι τοπικό και παραδοσιακό, αν θέλουμε να εναγκαλίσουμε τα ωφέλη της ηθαγένειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ανεμαρία. Όπως έλεγα και εγώ στην εισαγωγή μου ότι η ηθαγένεια δεν είναι αυτόνομη της υπηκότητας, ε, της εθνικής ηθαγένεια. ίσα ίσα είναι ένας τρόπος να την ε, προβάλλουμε, να της προσδώσουμε αξία. Ε, το, η πολυπολιτισμικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική. Κυρία μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω γαλλικά. Κατρίν Κισετζιάν, θα μιλήσω σήμερα το απόγευμα ε, αλλά νομίζω ότι θα ήθελα να πω κάτι τώρα το οποίο έχει σχέση με τη συζήτηση που κάνουμε τώρα. Ε, ακούστηκε σήμερα το πρωί, αλλά νομίζω ότι είναι θεμελιώδες και θα ήθελα να επιμείνω στο γεγονός ότι πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ των θεμάτων που έχουν άμεση σχέση με την ευρωπαϊκή ηθαγένεια ως ε, νέα στοιχεία της συνθήκης του Μάστριχτ και των οικονομικών δικαιωμάτων που έχουμε όλοι και τον αν είμαστε πολίτες ή όχι ε, δεν έχουν καμία σημασία. Έχουμε όλοι οικονομικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από την αρχική συνθήκη της Ρώμης και για τα οποία νομίζω ότι δεν υπάρχει ανάγκη για νέα νομοθεσία. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι καλύτερες πρακτικές, βέλτιστες πρακτικές, τις οποίες θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε καλύτερα και που θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε, αλλά για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και εγώ είμαι νομικός, αλλά με ανησυχεί ιδιαίτερα αυτό το γεγονός της ισόρευσης της νομοθεσίας, στην οποία χαρονόμαστε ακόμα και εμείς. 47 σελίδες οδηγίες για εμά ως νομικούς είναι πολύ δύσκολο να τη διαβάσουμε και την κατανοήσουμε, πολλό δε μάλλον για κάποιον ο οποίος δεν έχει νομικές γνώσεις, είναι σχεδόν αδύνατον. Και μια δεύτερη παρατήρηση, ε, να πω ότι με εξέπληξε η δεν με εξέπληξε το γεγονός ότι δεν ακούσαμε το τι μπορούμε να κάνουμε να επιλύσουμε κάτι πριν φτάσουμε στο δικαστή. Ο δικαστής είναι μια ιδιαίτερα δαπανηρή υπόθεση. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν όλες τις εναλλακτικέ δυνατότητες πρόληψης της ε, ε, επίλυσης διαφορών στο δικαστήριο. χρησιμοποίησα το Solvit, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Εδώ και 20 χρόνια το χρησιμοποιούσα. Δεν έχω δει τα στατιστικά στοιχεία, αλλά τότε που ασχολούμουν εγώ, περίπου το 80 με 85% των περιπτώσεων που έφταναν στο Solvit ε, επιλύονταν ε, πριν να φτάσουμε σε κανονική επίλυση διαφορών. Καλό είναι λοιπόν να χρησιμοποιούμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα και να μην προσπαθούμε να συσσωρεύουμε νόμου οι οποίοι θα είναι ει βάρο μα τελικώ. Ευχαριστώ. Συμφωνούμε απολύτως με αυτά που είπατε βεβαίως. Άλλη μία ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Παπαχριστόπουλος ονομάζομαι. Είμαι ο πρόεδρος ε, μιας ε, διεθνούς ένωσης ε, μη κυβερνητικής. Ευρωπαίοι σε όλο τον κόσμο. Europeans throughout the world. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο δεν ελήφθη υπόψη. Μιλάω για 35 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξακολουθούν να είναι Ευρωπαίοι πολίτες και πάρα πολύ λίγη δράση αναλαμβάνεται για αυτούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκτός ε, από την προξενική προστασία την οποία την εγκρίναμε και βεβαίως πολλά ε, μένει ακόμη να γίνουν ε, για το θέμα αυτό. Δεν έχει ληφθεί ιδιαίτερη δράση για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι άμα το σκεφτείτε θα μπορούσαν να αποτελούν μια ολόκληρη χώρα. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να ψηφίσουν ε, εύκολα στις ευρωεκλογέ και η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα είναι μια πάρα πολύ καλή ε, ιδέα γιατί θα διευκολύνει την συμμετοχή όχι μόνο εκείνων αλλά και άλλων ε, ε, Ευρωπαίων που ζουν Ευρωπαϊκής Ένωσης. νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να υπάρχει μια εκτελεστική υπηρεσία που θα ασχολείται ειδικά με τους ε, ανθρώπους που ζουν με τους ομογενείς πολίτες. Ε, έχουμε πάρα πολλές εκτελεστικές ε, υπηρεσίες που ασχολούνται με πολλά άλλα θέματα. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε το, ε, κάτι τέτοιο και για τους ανθρώπους αυτούς. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, για αυτήν την πολύ συγκεκριμένη προστασία, πρόταση. Συγγνώμη. Ο Μάικλ θέλει να τη σχολιάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για το, την ερώτηση αυτή. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν νομίζω με αυτό που είπατε και με αυτό που είπε και η Άννα Μαρία. Εν μέρη το πρόβλημα στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ότι η Ευρώπη εκπροσωπείται στα κράτη-μέλη συχνά ως το πρόβλημα και όχι ως η λύση. Έτσι αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στις περισσότερες περιπτώσεις όταν γίνεται νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο ε, ούτως ή άλλως πάντοτε ε, κατα, καταγράφουμε τις ψηφοφορίες, τον αριθμό των ψήφων, αλλά οι πολίτες δεν γνωρίζουν πώς οι, οι υπουργοί τους, από τα κράτη-μέλη, από τις ε, ε, κυβερνήσεις τους, τι ψήφισαν, τι παραχωρήσεις έκαναν, τι αποφάσισαν. Και πρέπει να καθησυχάζουμε τον κόσμο ότι το να είναι κανείς Βρετανός ή Σουηδός δεν αντικρούει την ιδέα της ευρωπαϊκής ηθαγένειας οι πολίτες στα κράτη-μέλη αυτά πρέπει να γνωρίζουν επακριβώς πώς ε, ε, συζητούν πώς ψηφίζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι υπουργοί τους και τότε είναι υπόλογοι, όχι όπως πιστεύουν κάποιοι πολίτες μόνο στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά πρέπει να είναι υπόλογοι και στα εθνικά κοινοβούλια και είναι υπόλογοι και στους πολίτες τους όταν ψηφίζουν. Αν λοιπόν δεν καλύψουμε αυτό το ε, δημοκρατικό έλλειμμα, τότε η υποστήριξη για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια θα μεωθεί. Για το θέμα της όλο και περισσότερης νομοθεσίας, εγώ είμαι υπέρμαχος του ότι όσο μεγαλύτερη είναι μια, ενώ όσο μεγαλύτερος είναι ένας, μεγάλος οργανισμός, τόσο καλύτερος πρέπει να είναι ο απολογισμός των πόσων των πραγμάτων πρέπει να κάνουμε περισσότερο και αυτών πρέπει να κάνουμε λιγότερο. Και δεν έχουμε κάνει κάτι τέτοιο και πρέπει να το κάνουμε. Αν θέλουμε λιγότερους νόμους, τότε ο τρόπος να το πετύχουμε αυτό είναι να έχουμε ανοιχτές συζητήσεις μεταξύ των ε, κοινοβουλίων στα οποία νομοθετούμε και με το Συμβούλιο των Υπουργών για να ε, δούμε τι γίνεται, γιατί σε αυτό το επίπεδο λαμβάνεται η απόφαση για την ομοθεσία. Δεν επιβάλλεται τίποτε όπως νομίζουν ε, οι Βρετανοί, όπως νομίζουν άλλοι ε, ακροδεξιοί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώς προτείνει αν οι συνομοθέτες δεν το δεχθούν και δεν ε, συμφωνήσουν, ε, ε καταραίει η πρόταση αυτή πηγαίνετε ε, στο Μπέρμιγχαμ, στο Μπρίστολ, ε, στο ε, Αμβούργο, στο δρόμο και ρωτήστε έναν πολίτη πού πιστεύουν ότι βρίσκεται η εξουσία. Οι περισσότεροι από αυτούς θα σας πούν ότι οι δικές τους κυβερνήσεις έχουν πάρα πολύ μικρή εξουσία όσον αφορά τις Βρυξέλλες. Και αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, ε, όλα αυτά για τα οποία συζητούμε σήμερα, σε 10 χρόνια πάλι ακόμα θα τα συζητάμε, γιατί όσο μεγαλώνει η οικονομική κρίση, οι άνθρωποι και κυρίως ε, στα ακραία κόμματα ψάχνουν κάτι ή κάποιον να κατηγορήσουν. Και είτε, είτε η Ευρώπη θα είναι ή ένας μεμονωμένος άνθρωπος ο οποίος θεωρούν ότι ήρθε στη χώρα τους από μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα να σου πάρει τη δουλειά, το σπίτι, τις υπηρεσίες, Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να συζητήσουμε τα ωφέλη του να είμαστε ε, πατριώτες, περήφανοι, αλλά να είμαστε και Ευρωπαίοι πατριώτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μάικολ. Πράγματι, ακόμα και αν δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε σε κάθε ε, Ευρωπαίο πολίτη να ε, κάνει μια αναφορά στην Ευρώπη για μια ερώτηση για να έχει ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, από τη συζήτηση φαίνεται ότι η ενημέρωση ε, μέσω πρόληψης, μέσω του Solvit, μέσω του Ευρωπαίου Μεσολαβητή, θα πρέπει να ενισχυθεί, να ξέρουν οι πολίτες ποιοι είναι. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως έχει ανοιχτές συζητήσεις, Μάικολ, ε, αναμεταδίδονται στο διαδίκτυο, πολύ συχνά ξέρουμε τι ψηφίζει ο κάθε Ευρω... Ευρωβουλευτής. Υπάρχει αρκετή διαφάνεια λοιπόν σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα να το επενθυμίσω αυτό και να το επισημάνω, διότι δεν ισχύει παντού. Ο κύριος, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Hans Modern από την πλατφόρμα των πολιτών που συνήθως αυτό που κάνουμε είναι να ενημερώνουμε για την Ευρώπη. Βλέπω εδώ στην αίθουσα εκπροσώπους από διάφορες οργανώσεις τις οποίους γνωρίζω τις περισσότερες φορές ε, και τους ευρωβουλευτές φυσικά. Εσείς γνωρίζετε τους ευρωβουλευτές ε, και ο κόσμος σας γνωρίζει. Το θέμα είναι όμως ότι όταν μιλάμε με πολίτες εκτός της ευρωπαϊκής ε, φούσκας, αυτοί δεν ενδιαφέρονται για την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν έχει σημασία για αυτούς. Θέλουν να ξέρουν τι είναι καλό για αυτούς και θέλουν να τους ε, διαβιβάζονται αυτά τα πράγματα με τέτοιο τρόπο ώστε να τους ενημερώνουν με σύντομο και ωραίο τρόπο. Και αυτό που κάνουμε εμείς τις περισσότερες φορές όταν διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτά που αναρτούν οι περισσότεροι ε, είναι ότι είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν είναι ευχάριστο, δεν διαβάζεται με ευχάριστο τρόπο και είναι και ιδιαίτερα δυσνόητο εάν κάποιο δεν έχει ένα πτυχίο και είναι μάλλον ανιαρό αυτό που διαβάζει. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε λοιπόν και πρέπει να αλλάξει είναι ε, τον επόμενο 1,5 χρόνο να δούμε με ποιο τρόπο διαβιβάζουμε αυτό που διαβιβάζουμε. Πριν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα εξηγήσουμε στον κόσμο πόσο καλύτερη είναι η ζωή τους, θα πρέπει ίσως να σκεφτούμε με ποιο τρόπο θα πρέπει να επικοινωνούμε. Και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι η λύση, είναι ένα εργαλείο. Το ραδιόφωνο είναι εξίσου σημαντικό, όπως είναι και η τηλεόραση, και ιδίω όταν αναφερόμαστε σε διάφορε ε, ηλικιακέ ομάδε, εκεί διαφοροποιείται ο τρόπο με ε, τον οποίο διαβιβάζουμε ένα μήνυμα και ε, πώ επικοινωνεί ο καθένα. Και θα πρέπει να το σκεφτούμε όλοι αυτό, όχι μόνο οι Ευρωβουλευτέ, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι όσοι είμαστε εδώ παρόντε, διότι οι περισσότεροι γνωρίζουμε τι δουλειά κάνει ο καθένα. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σα. Συμφωνούμε απολύτως με την παρέμβασή σας. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε είναι πολύ σημαντικός ε, και η παιδαγωγική πτυχή θα πρέπει να ε, υπάρχει εδώ. Ε, εσείς λοιπόν που διαβιβάζετε και ασχολείστε με θέματα επικοινωνίας υπάρχουν διάφοροι τρόποι επικοινωνίας ακόμα και για μικρά παιδιά. Ε, είναι θέμα ε, του πώς διαβιβάζετε τι. Στην περιοχή μου για παράδειγμα υπάρχει ε, ένας χώρος που λέγεται Amphorop που επιτρέπει να επικοινωνούν, μπορούν οι ευρωβουλευτές να πάνε σε σχολεία, σε ηλικία, σε δημοτικά για να δουν τι γίνεται. Ε, δυστυχώς δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο και πολύ γνωστό αυτό. Ε, αναφερθήκατε και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός. Ε, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα αντίβαρο, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό στις χώρες μας. Η εθνική πολιτική τάξη. Και πολύ συχνά αυτή η εθνική πολιτική τάξη ε, που ε, είναι ανοιχτή προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εισακούγεται πολύ περισσότερο από τους ε, ευρωβουλευτές έχει ένα, μια τάση να υποβαθμίζει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα παρουσιάζει ως έναν επίτροπο, κάτι πολύ περίπλοκο, μια νομοθεσία που είναι πολύ δυσνόητη και κυρίως πλήττουν τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και σε επίπεδο εθνικής πολιτικής τάξης, σε όλα τα κόμματα, σε όλες τις πολιτικές οικογένειες και θα πρέπει ε, αντιθέτως να είναι μια πολύ σημαντική συνιστόσα, πολύ πιο σημαντική και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για τον τρόπο με τον οποίο ανταλαμβανόμαστε την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Θέλετε να απαντήσετε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Συμφωνώ μαζί σας ε, για τα περισσότερα. Το θέμα είναι ότι για τον επόμενο 1,5 χρόνο είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχουν μόνο οι κακές Βρυξέλλες εντό εισαγωγικών. Θα πρέπει αυτό να γίνει αντιληπτό σε τοπικό επίπεδο, γιατί είναι αυτό το επίπεδο το οποίο μετράει για, τους πολι... για... για όλους μας και επίση θα πρέπει να υπάρχει πολύ περισσότερη επικοινωνία επιτόπου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει infopoint ε, στην ε, πόλη κάθε δύο εβδομάδε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Θα πρέπει να γίνεται με ευχάριστο τρόπο, διασκεδαστικό, να ε, συγκεντρώνεται ο κόσμο και να μπορεί να θέσει ερωτήσει, οι οποίε τι περισσότερε φορέ δεν θα είναι πολύ συγκεκριμένε. Ε, μπορεί να θέλουν γιατί, να ξέρουν γιατί η Βρυξέλλε έχει τόσου πολλού γραφειοκράτε. Και δεν είναι σωστή απάντηση ότι έχει 55.000 μόνο υπαλλήλου που είναι λιγότεροι από, τις, από όσους έχει ο Δήμος του Μπέρμιγχαμ, θα πρέπει να του απαντάτε με τρόπο ώστε να σας κατανοούν και να κατανοούν ότι ε, ζείτε και εσείς τη ζωή σας στο ίδιο επίπεδο. Και δεν έχει σχέση με την ευφυή αυτό, απλώς ε, είναι το γεγονός ότι ο κόσμος ζει τη ζωή του, δεν ζει εδώ στις Βρυξέλλες και θα πρέπει λοιπόν να περάσουμε ε, σε απλούς κανόνες και να μιλούμε στους πολίτες, να τους αφήνουμε να θέτουν ερωτήσεις, ε, για παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο διαβιβάζονται κάποια από τα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει χρησιμότητα ε, εάν δεν επιτρέπετε τις επικρίσεις ε, γιατί θεωρείτε ότι θα αποτύχετε. Πρέπει να αποτύχετε γιατί και αυτό μέσα στη ζωή είναι. Φρανκ ε, Μπένιον Frank Από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρωτοβουλία που αναλάβατε. Είναι μια κοινή πρωτοβουλία ε, και θα επανέλθω σε αυτήν. Σήμερα όλοι μιλάμε για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Αλλά όπως είπε και Άλισον Μακδόνελ, η έννοια αυτή είναι πολύ ασαφή στις συνθήκες, διότι αναφέρεται σε κυρίαρχα κράτη, αναφέρεται σε θέματα φορολόγησης, αναφέρεται σε θέματα εκπαίδευσης, τα οποία δεν, στα οποία δεν μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν ε, σαφώς περιορίζεται η έννοια ε, της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Τώρα το άρθρο 20 της ε, συνθήκης ε, αναφέρεται στην ελεύθερη κυκλοφορία και στο δικαίωμα παραμονής και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα είπαμε, τα αναφέραμε σήμερα το πρωί, αλλά αυτά τα δικαιώματα αφορούν 3 με 4% του συνολικού πληθυσμού. Ένα δεύτερο στοιχείο στο άρθρο 20 είναι το δικαίωμα ψήφου, το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα συζητήσουμε το απόγευμα. Αλλά το άρθρο 20 λέει ότι αυτά τα δικαιώματα μεταξύ άλλων, μεταξύ άλλων. Άρα τι σημαίνει αυτό το μεταξύ άλλων, τι περιέχει η κυρία Ρέντιν στην παρέμβασή της στην Επιτροπή Περιφερειών τον Νοέμβριο είπε ότι πολλοί πολίτες ε, περιμένουν συγκεκριμένα αποτελέσματα από την Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχω δει σε κανένα έγγραφο, σε καμία τεκμηρίωση μία συγκεκριμένη αναφορά στα δικαιώματα, ενώ χειροπιαστά ατομικά δικαιώματα τα οποία είναι εφαρμόσιμα. Δεν έχω δει έναν κατάλογο πουθενά. Και την τελευταία δεκαετία σε διάφορους τομούς, τομείς έχουν εδρεωθεί δικαιώματα. Παραδείγματο χάρη στην, στις αερομεταφορές η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικαίωμα σε κάθε πολίτη, ε, το δικαίωμα της αποζημίωσης όταν υπάρχουν ε, προβλήματα στο ταξίδι του. και λέει ότι μπορεί να πολεμήσει για τα δικαιώματά του αυτά στα εθνικά δικαστήρια και υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις. Στις τηλεπικοινωνίες υπάρχει, υπάρχουν όλες διαδικασίες για την περιαγωγή, το roaming ε, και έχουμε και εκεί δει πάρα πολλές ε, περιπτώσεις προσφυγών ε, όσον αφορά και την, τα δικαιώματα μεταφοράς στην κινητή τηλεφωνία. Αλλά και στον τομέα της υγείας υπάρχουν, έχει επιτευχθεί πρόοδος δεδομένου ότι μπορούν Ευρωπαίοι πολίτες σε μια χώρα να ε, χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίε υγείας σε μια άλλη χώρα. Αυτές, αυτά τα δικαιώματα έχουν εδρεωθεί, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να είναι διασυνοριακά. Ε, δεδομένου ότι ένας Ευρωπαίος πολίτης που μένει σε μια χώρα, στη χώρα του και βλέπει το λογαριασμό της κινητής τηλεφωνίας του, διαπιστώνει ότι το κόστος ας πούμε έχει κατέβει. Και πάλι Αυτά τα οποία εμείς θέλουμε να εδραιώσουμε είναι την ισοτιμία των δικαιωμάτων μεταξύ ενός πολίτη και ενός άλλου. Δηλαδή μεταξύ ενός που χρησιμοποιεί ένα αεροπλάνο και του άλλου που χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο. Έτσι ώστε και οι δύο να χαίρουν των ιδίων δικαιωμάτων εφόσον είναι Ευρωπαίοι πολίτες και έχουν την ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Εδώ σήμερα βλέπουμε ε, το Κοινοβούλιο και το, την Κομισιόν, δύο βασικούς παίκτες και αυτοί πρέπει να συνεργάζονται. Εάν κανείς πάει στο Ζάβεντεμ βλέπει τα δικαιώματα των ταξιδιωτών κολλημένα στον τοίχο και από κάτω λέει Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εν συνεχεία βλέπει μία άλλη αφίσα και από κάτω λέει Ευρωπαϊκή Εκτελεστική Επιτροπή, Κομισιόν αυτά δεν μπορούν να συγκεραστούν, δεν μπορούν να ενωθούν. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να χειριστούμε τα θέματα ξεχωριστά μία εβδομάδα να ασχοληθούμε με τον τομέα της υγείας και εκεί να επικεντρώσουμε την παρουσίαση των, ε, της Ευρωπαϊκής Ιθαγέννης και των Δικαιωμάτων και την άλλη εβδομάδα oh, να μιλήσουμε για άλλους τομείς. Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ε, κύριε, έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, προέρχομαι από το Düsseldorf της Γερμανίας και θέλω κι εγώ να σχολιάσω αυτά που είπε ο κύριος εκεί πίσω για την Ευρώπη των πολιτών. Πριν από δύο εβδομάδες περίπου ο Αμερικανός Πρόεδρος ε, έκανε την ομιλία του για το State of the Union, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τη χώρα του και την κατάσταση και είπε προς τον πρόεδρο του Κογκρέσου και τα μέλη του, είπε «Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, αγαπητοί πολίτες, dear citizens, αν κοιτάξτε και την ετήσια ομιλία του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κομισιόν του κυρίου Μπαρόζου, η ομιλία του αρχίζει ως εξής. Κύριε Πρόεδρε, ε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, τελεία και παύλα. Για συμπολίτε ούτε νίξη δεν γίνεται. Καμία αναφορά. Και μου φαίνεται ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα του τι δεν πάει καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολλά τέτοια παραδείγματα υπάρχουν και όλοι μπορούμε στην αίθουσα αυτή να αναφέρουμε μερικά. Παραδείγματο χάρη το πρόγραμμα εργασίας ε, της ε, Ευρωπαϊκής Προεδρίας του Συμβουλίου όπως ας πούμε αηφορία, δημοσιονομική σταθερότητα, ασφάλεια κλπ. κλπ. Πολίτες, που, το, πολίτες, το θέμα πολίτες, πού βρίσκεται. Το θέμα αυτό είναι συνήθως χωμένο σε κάποια ατζέντα στα χαμηλά, πίσω-πίσω. Η προσωπική μου άποψη δεδομένου ότι προεδρεύω μιας μικρής ένωσης στο Düsseldorf που ασχολείται με την διάδοση του ευρωπαϊκού μηνύματος. Το μήνυμα μου λοιπόν είναι ότι όταν γίνονται ό,τι γίνεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εννοούν ότι γίνονται για τον πολίτη. Γίνονται για την παγίωση ενός εξαιρετικά περίπλοκου νομικού καθεστώτος. Εδώ μιλάμε για νομοθεσία, για ένα οικοδόμημα νομοθετικό, κανονιστικό, όχι για ένα οικοδόμημα του πολίτη. Όταν μιλάμε όμως για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να περιορίζουμε το οικοδόμημα αυτό σε νομικιστικές, δικαστικές, δικονομικές και κανονιστικές ρυθμίσεις. Αυτά είναι νεκρά, ε, ε, νεκρές πτυχές, ε, πτυχές χωρίς ψυχή. Εμείς θέλουμε να δώσουμε σώμα και ψυχή στο οικοδόμημα αυτό. Και το σώμα και η ψυχή είναι οι πολίτες, οι άνθρωποι. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια έκκληση, επιτρέψτε και σε μας να συζητήσουμε και να προβάλλουμε τα πράγματα που μας αφορούν πέραν όλων αυτών των παγιωμένων νομικών και κανονιστικών διατάξεων. Και επίσης θέλουμε μια φορά επιτέλους ο πρόεδρος της Ευρώπης να συμπεριλάβει στην προσφώνησή του και εμάς, τους πολίτες και το λέω απευθύνουμε κυρίως στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Πιστεύω ότι αυτό θα δώσει ένα σαφές μήνυμα. Είναι πολύ σημαντικό να μας συμπεριλάβει για να δει, για να καταλάβουμε κι εμείς ότι εννοεί εμάς, ότι απευθύνεται σε εμάς. Διαφορετικά για, ποιο, για ποια δημοκρατία μιλάμε και για ποιο έτος των πολιτών. Είναι είναι σαν να λέει κάποιος διευθυντής ενός ζωολογικού κήπου ότι φέτος ε, θα ονομάσουμε το, το έτος μας το έτος των ζώων. Ε, μα αυτονόητο δεν είναι αυτό. Για μας δεν μιλάει, σε μας δεν απευθύνεται. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε το κέντρο αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είμαστε ε, χωμένοι κάπου στα, στα, στα πάνω στο ράφι να πούμε να σκονιζόμαστε και να μην μας λαμβάνουν υπόψη. Ευχαριστώ πολύ, ναι. Πράγματι. Ενδεχομένω ο κύριο Νέμιτ ε, να μπορεί να σα πει ορισμένα πράγματα για αυτό που είπατε σε σχέση με τον κύριο Παρόσο. Όμω ε, η μεταφορά που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω είναι σαν ένας μεγάλος ε, καθηγητής ιατρικής γνώριζε το, την ε, περίπτωση του κάθε ασθενή. Ε, κάπως έτσι θα το παρουσίαζα. Ευχαριστώ πολύ. Νίκολας Νιωμάν, είμαι Γενικός Διευθυντής ε, της οργάνωσης που παρουσίασε ήδη ο κύριος Παπαχριστόπουλος, Europeans Throughout the World. Εμείς συνεργαζόμαστε με πολλές έχουμε ως μέλη πολλές ενώσεις ε, αποδήμων ε, που ζουν σε άλλες χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αλλά και απόδημους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά προβλήματα έχουν επιληθεί στο πλαίσιο των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως εξακολουθούν να υφίστανται εκτός αυτών. Και αντίθετα με αυτό που είπε προηγουμένως η κυρία Βαλεάν, υπάρχουν ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάνουν διακρίσεις ε, μεταξύ των ε, πολιτών του και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα από αυτά. Συνταξιούχοι που είναι Ευρωπαίοι πολίτες, σας υπενθυμίζω, αν φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο ή φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ζήσουν αλλού στον κόσμο, ε, βλέπουν τις συντάξεις τους να παγώνουν ε, ε, στο επίπεδο στο οποίο ήταν τη στιγμή που μετανάστευσαν. Είναι όμως Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτό μπορεί να έχει πολύ αντίξω αποτέλεσμα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια συγκεκριμένη περίπτωση που είδα προσφάτως. Κάποιο γύρισε από την Αυστραλία υπήρξε, υπήρχε παλιά συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Αυστραλίας, όμως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα opt-out που περιορίζει τη δυνατότητα των, συνταξιο, των συνταξιούχων να ε, μετακινούνται, να ταξιδεύουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν βγει έξω από το Ηνωμένο Βασίλειο, χάνει την ε, αγγλική του σύνταξη. Είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι παράνομο, όμως τα βρεκανικά δικαστήρια ε, δικαίωσαν την πρακτική αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οργανώσεις ε, που εκπροσωπούν αυτούς τους ανθρώπους που είναι από 35 έως 60 εκατομμύρια ανάλογα με τις περιπτώσεις, ανάλογα με το κατά πόσο λαμβάνουμε υπόψη όσο έχουν διπλή υπηκότητα ή πολλαπλή υπηκότητα. Όταν έχει κανείς διπλή υπηκότητα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μικρότερο το πρόβλημα. Αν κάποιος όμως ε, μεταναστεύσει στον Καναδά για παράδειγμα ε, για να μπορεί να έχει πρόσβαση ε, σε κάποιες θέσεις απασχόλησης πρέπει να γίνει Καναδός. Αν όμως με το να γίνει Καναδός χάνει την ε, ευρωπαϊκή του υπηκότητα που συμβαίνει σε μερικές χώρες αλλά όχι σε όλες ευτυχώς, αυτό μπορεί να έχει πολύ σημαντικές συνέπειες. Σήμερα το απόγευμα θα αφιερώσουμε το χρόνο μας στα στο δικαίωμα ψήφου. Δεν θέλω να πω σε πολλέ λεπτομέρειε για την ώρα, αλλά θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν διακρίσει κατά Ευρωπαίων πολιτών που ζουν εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, όταν έχουν λυθεί τα προβλήματα ε, στη, Ένωση, Ευρωπαϊκής Νομίζω ότι επιτέλου πρέπει να κάνουμε και κάτι ε, για όσου βρίσκονται εκτό. Ευχαριστούμε που θέτετε αυτό το θέμα, το πολύ συγκεκριμένο των αποδήμων εκτό και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλετε να πάρετε το λόγο κύριε Νέμιτ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα της ηθαγένειας, την έννοια της ηθαγένειας, δεν είναι απλώς ε, νο, νομικός και δεν ε, εξαντλείται στον τίτλο 5 της συνθήκης, μόνο δηλαδή στο κεφάλαιο περί ηθαγένειας. Αν δείτε την έκθεση περί ηθαγένειας του 2010, θα δείτε και πάλι, θα το δείτε και ε, στην επόμενη έκθεση που θα δημοσιευθεί το Μάιο, Μιλάμε για 25 δράσεις που συμπεριλαμβάνουν που πηγαίνουν πολύ πέρα από το κεφάλαιο περί ηθαγένειας. Είναι γεγονός ότι η έννοια της ηθαγένειας ε, όταν ε, το βλέπουμε υπό καθαρά νομικό πρίσμα είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Ε, είναι γεγονός ότι στο πλαίσιο της έκθεσης προσπαθούμε να δούμε θέματα που είναι ε, μεγάλου ενδιαφέροντος για συγκεκριμένους ε, πολίτες ε, στο επίπεδο, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης. Δεν είναι όμως μια νομικήστικη προσέγγιση η οποία περιορίζεται μόνο στα, στο κεφάλαιο περιθαγένειας. Για το δεύτερο θέμα που ετέθη, και εγώ το, είπα, το είδα το, το πρόσεξα αυτό σε σχέση με το, την κατάσταση της Ένωσης, αλλά να είμαστε δίκαιοι, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε πει ένα πολύ σημαντικό πράγμα στην ίδια ομιλία, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι στην επό, επόμενες ευρωεκλογές ε, πρέπει ο υποψήφιος της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, πρέπει να είναι γνωστός στον κόσμο από τις πολιτικές ομάδες. Εντάξει, δεν προτείνουμε άμεση βέβαια εκλογή του Προέδρου όπως συμβαίνει στις Ηνωμένε Πολιτείε. όμως νομίζω ότι είναι ε, πραγματικά ε, μεγάλο, ε, μεγάλο μέλημα ε, και του Προέδρου και της Αντιπροέδρου να δώσει με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερο βάρος στην, ε, στο συγκεκριμένο ε, τίτλο. Καταλαβαίνω λοιπόν τι είπατε και το σημειώνω, αλλά θα ήθελα να επενθυμίσω ότι η συγκεκριμένη Επιτροπή στη σύνθεσή της στην τρέχουσα, ο κύριος Μπαρόζο και η κυρία Ρέντινγκ, η Αντιπρόεδρος, ε, προσπαθούν να εφαρμόσουν κάτι που το έχουμε πολλές φορές πει στο παρελθόν, ελπίζω όμως αυτή τη φορά όντως να συμβεί και πιστεύουμε, εγώ τουλάχιστον πιστεύω, ότι τα κόμματα που θα το κάνουν αυτό θα έχουν ένα μεγάλο ε, πλεονέκτημα και θα έπρεπε να επιβραβευτούμε περισσότερες ψήφους ε, ε, όταν πούν ποιος είναι ο δικός τους υποψήφιος για το χρήσμα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νέμιτς. Ευχαριστώ πολύ. Εργάζομαι για το Air Center, μια μη κυβερνητική οργάνωση στο Λονδίνο και είμαι και μέλος της ε, Συμμαχίας του Ηνωμένου Βασιλείου για τους Ευρωπαίους Πολίτες. Και θα ήθελα να απαντήσω σε κάτι το οποίο ανέφερε ο κύριος από τον Τίλσεντορ και το οποίο χρονοκρότησαν όλοι. Διότι νομίζω ότι η ιδέα μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που είναι πολύ σημαντική ε, δεν ε, είναι το απαραίτητο για αυτούς που είναι εδώ σήμερα. Αυτό που ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους πολίτες είναι τα καθημερινά δικαιώματα και η πρόσβαση σε αυτά. Θα αναφερθώ σε κάποια θέματα τα οποία αναφέρθηκα σήμερα ως προβλήματα της μεσαίας τάξης. Ε, είμαι λίγο διαφιλονικούμενο το ζήτημα, επίμαχο, αλλά τον περισσότερο κόσμο τον ενδιαφέρει να αγοράσει αυτοκίνητο, να πληρώσει το λογαριασμό του, τηλεφώνου του. Ε, οι άνθρωποι με τους οποίους έρχομαι σε επαφή εγώ έχουν πιο βασικές ανάγκες που φαίνεται να τις αγνοούμε και νομίζω ότι και εσείς εδώ τις αγνοείτε. Το βασικότερο θέμα το οποίο αντιμετωπίζω καθημερινά ε, έχει να κάνει με ε, ε, υπηκόους της οχο που είναι είτε Ρωμά είτε άστεγοι και έχουν προβλήματα τα οποία δεν έχουν σχέση μόνο με καλή διοίκηση. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και δελεαστικό, αλλά αφορά την καθημερινότητά τους και μάλιστα με πολύ σοβαρά προβλήματα. Όταν ε, προσπαθείς πούμε να μιλήσεις με μια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία δεν αναγνωρίζει καν ε, τη χώρα σου ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσβαση σε έγγραφα επίσης. Το γεγονός ότι η οδηγία για την Ευρωπαϊκή Φυγένεια θέτει ένα όριο έξι μηνών ή τουλάχιστον αυτό έχω αντιμετωπίσει εγώ καθημερινά. Ε, αυτό το εξάμεινο συνήθως περνάει ε, με τα όσα πρέπει να κάνει η υπηρεσία συνόρων. Υπάρχει ε, μια περίπτωση ε, ενός ανθρώπου ε, με τον οποίο ασχολούμαι, ο οποίος είναι μέλος μιας χώρας σε ΟΚ και το διαβατήριό του το έχει κατασχέσει στην πραγματικότητα η υπηρεσία των τελωνίων για τρία χρόνια και δεν έχει πρόσβαση ε, σε τίποτα ε, και η ζωή της είναι πάρα πολύ δύσκολη λόγω ε, απίστευτων καθυστερήσεων στην επίλυση της υπόθεσής της. Υπάρχουν επίσης και κάποιοι φραγμοί οι οποίοι τίθενται από τις εθνικές αρχές για πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα και αναφέρομαι σε αυτό συγκεκριμένα διότι αυτό είναι ο τομέας με τον οποίο ασχολούμαι εγώ. Αλλά για παράδειγμα, ο αριθμός εθνικής ασφάλισης, ο ΆΜΚΑ στην Ελλάδα. Ε, το τι γίνεται με αυτού του ανθρώπου στο Ηνωμένο Βασίλειο και αν δεν μπορούν να έχουν ένα τέτοιο αριθμό και δεν έχουν κοινωνικά επιδόματα. Λυπάμαι που έφυγε ο κύριο Κάσμαν διότι αναφέρθηκε σε μια κοινωνία και ε, ότι ένδειξη κοινωνία και του πολιτισμού είναι ο τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στι μειονότητε. Έχει σημασία όμω να συνεργαζόμαστε και με τι τοπικέ αρχέ. και θα ήθελα να το πούμε λίγο σαφέστερα. Ε, θα εκπαιδεύσουμε του ανθρώπου που ε, εργάζονται στι τοπικέ αυτοδιοικήσει για να επιλύουν τα προβλήματα καλύτερα ή αναφερόμαστε σε επίλυση διαφορών. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε κάτι ενδιάμεσο. Δεν πρέπει απαραίτητο να έχουμε διαδικασία σε επιπαραβάση ή κάτι αυτή τη κλίμακτη. Νομίζω ο κύριο Μακουίν αναφέρθηκε στην αδυναμία των πολιτών απέναντι στι δομέ. Δεν πρέπει απαραίτητο να φτάσουμε σε διαδικασία επί για να έχει κάποιο πρόσβαση στα δικαιώματά του. Αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να βασιζόμαστε και σε αποφάσει καλή πίστη. Ε, υπάρχει ένα μεγάλο κοινό λοιπόν μεταξύ των δικαιωμάτων και της πρόσβασης σε αυτά και θα ήθελα να ξέρω τι έχετε να πείτε. Πώς μπορούμε να ε, διαρθρώσουμε, να λύσουμε το τι γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Ε, τι γίνεται με τις αποφάσεις που πλήττουν ε, τους Ευρωπαίους πολίτες που μπορεί να μην εκπροσωπούνται εδώ σήμερα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κορατσαμπίλτ. Δεν έχω απάντηση να σας δώσω, αλλά ασχολούμαστε ιδιαίτερα ε, κυρίως σε θέματα ε, διακυβέρνησης ενιαίας αγοράς. Εμείς δεν εργαζόμαστε κατά των τοπικών αρχών ή σε επίλυση διαφορών με τις τοπικές αρχές. Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές, διότι ανήκουμε στην ίδια κοινωνία ε, που έχει ως τελικό αποδέκτη τον πολίτη. Ε, και κανονικά από τις Βρυξέλλες θα έπρεπε να φτάνουμε σε οποιοδήποτε μικρό χωριό, σε οποιαδήποτε άκρη της Ευρώπης ε, και θα πρέπει να συνεργαζόμαστε καλύτερα και εκ των προτέρων. Και αυτό εγκρίναμε στην Ολομέλεια πριν από κάποιες εβδομάδες. Και εκ των προτέρων. Πώς θα φτάσει αυτό στην καθημερινότητά σας, στη δουλειά σας, στις σπουδές σας. Και νομίζω ότι πολύ συχνά είναι η ερμηνεία που είναι πολύ περιοριστική ή λιγότερο περιοριστική, ιδίω για τις οδηγίες τελικώ καταλήγουμε σε κάτι τελείω διαφορετικό. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Στη Σουηδία πριν από μία-δύο εβδομάδε υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα διότι δεν μπορούσαν ε, να αγοράσουν εισιτήριο μέσω SMS για το λεωφορείο. Το κόστο του εισιτηρίου είναι 3 ευρώ και αυτό προέκυψε από μία εφαρμογή μια οδηγία που στόχο είχε να διευκολύνει τι πληρωμέ και να τι ε, απλουστεύσει. Αλλά εγκρίθηκε σε εθνικό επίπεδο με τέτοιο τρόπο ώστε έθεσε μία σειρά από απαιτήσει να έχει κάποιο κάνει πρώτερη εγγραφή καταγραφεί και ούτω καθεξής. Και αυτό φυσικά ε, ήταν και ένα μέτρο καταπολέμησης τη νομιμοποίηση παρανόμων ε, εσόδων και νομίζω ότι τα 3 ευρώ του λοφορείου δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος να ξεπλύνει κάποιο χρήματα. Είναι ένα βλακώδες μικρό παράδειγμα το οποίο όμως δημιούργησε πολλά προβλήματα σε χιλιάδες ανθρώπους που πήγαιναν στη δουλειά του και δεν μπόρεσαν να αγοράσουν εισιτήριο στο λεωφορείο. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν να παρακολουθούμε πιο στενά και να συνεργαζόμαστε πολύ καλύτερα ακόμα και στην αρχή της νομοθετικής διαδικασίας με τα Εθνικά Κοινοβούλια και με τις τοπικές αρχές. Ε, οι Δήμοι στην Ευρώπη έχουν το 70% της δουλειά τους που προέρχεται από τις Βρυξέλλες. Έχουν λοιπόν κοινή ευθύνη στο τελικό αποτέλεσμα που είναι η βελτίωση της δικής σας της ζωής. Και αν δεν έρθει αυτό στην επιφάνεια και δεν συνεργαστούμε μαζί τους, ε, είναι, θα είναι πρόβλημα. Διότι εγώ πάντα στη Σουηδία ακούω ότι φταίει πάντα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και αν δεν σπάσει αυτό το ταμπού, όχι με επίλυση διαφοράς, αλλά μέσω συνεργασίας, για να έχουμε αποτελέσματα για τους πολίτες, δεν θα το επιτύχουμε μόνο από τις Βρυξέλλες. Είναι αδύνατον. Ε, επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμα. Γιατί οι άνθρωποι που εργάζονται σε εθνικούς φορείς ε, δεν αποκαλούνται ε, γραφειοκράτες, αλλά αποκαλούνται πολιτικοί σύμβολοι και όλοι όσοι δουλεύουν στις Βρυξέλλες είναι γραφειοκράτες. Όλοι δουλεύουμε για να εφαρμόσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εάν εσείς λοιπόν δεν αλλάξετε ε, αυτή την άποψη ότι ό,τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες είναι γραφειοκρατικό, κατά των πολιτών, κατά του λαού είναι τεχνοκρατικό και ό,τι συμβαίνει στη χώρα μας είναι καλό και είναι για τους πολίτες, ε, θα ε, είστε αυτοί που θα έχετε πρόβλημα, διότι εμείς είμαστε αδύναμοι χωρίς εσάς. Όλοι εμείς ε, ε, σας έχουμε εδώ σήμερα γιατί σας καλέσαμε. Θέλουμε να ακούσουμε και άλλους ανθρώπους. Δεν θέλουμε μόνο πολιτικούς και τεχνοκράτες. Δεν θα ήσασταν εδώ σήμερα αν δεν θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Θα σας δώσω το λόγο αμέσως μετά, αλλά έχει ζητήσει να απαντήσει και ο κύριος Νέμιτς. Uh, Πολύ σύντομα. Να απαντήσω στην κυρία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Βεβαίως, πρέπει να έχουμε όλα αυτά τα μέσα που αναφέρεται. Διαδικασίες ε, προσφυγής σε περίπτωση παραβιάσεων, αυτό δεν, έχει επιπλέον κόστος για την Κομισιόν και στον Ηνωμένο Βασίλειο για αυτά που είπατε έχουμε μια διαδικασία προσφυγής που αφορά όχι αποκλειστικά αλλά κυρίως επικεντρώνεται σε ε, υπηκόους από τη Βουλγαρία και την κοινότητα των Ρωμά πρέπει να εξηγήσουμε πολλές φορές στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους Δήμους ότι δεν εξυπηρετεί σε τίποτα η πολιτική της παρεμπόδισης των προσκομμάτων, η αρνητική αντιμετώπιση κλπ. Αυτά δεν είναι καλά, δεν ωφελούν σε τίποτα. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας όφελος δεν υπάρχει. Πρέπει λοιπόν να τους πείσουμε ότι ε, δεν πρέπει να παρουσιάζουν προσκόμματα. Όμως ε, στις περιπτώσεις που είναι αμετάκλητοι και δεν αλλάζουν τη στάση τους πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία κυρώσεων, τη διαδικασία προσφυγής εναντίον τους. Ε, δεν μπορώ όμως να πω, εγώ δεν ισχυρίζουμε ότι όλες οι επιτυχίες προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Εγώ πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας ε, υλοποίηση των διατάξεων ε, οφείλεται στους ήρωες εθνικούς δικαστές οι οποίοι εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία. Και οργανισμοί και ενώσεις σαν τις δικές σας ε, δίνουν, προσφέρουν ακριβώς αυτή τη δυνατότητα ενημέρωση στους πολίτες, να χρησιμοποιούν τα καλύτερα μέσα σε περίπτωση που πρέπει να ε, δράσουν ή να προσφύγουν. Η κυρία Βάλεαν και εγώ ήθελα να πω ότι ε, το θέμα εδώ δεν είναι η ε, εφαρμογή της αρχής επικουρικότητας και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Όταν μιλάμε εμείς εδώ για ευρωπαϊκή ηθαγένεια, δεν θα πρέπει να την ερμηνεύουμε ως ηθαγένεια βρυξελιώτικη, δηλαδή ότι είναι, αφορά μόνο τους ε, κοινοτικούς ε, ε, πολίτες που βρίσκονται στις Βρυξέλλες. Δεν περιορίζεται τοπικά η έννοια. Η ευρωπαϊκή ηθαγένεια αφορά όλους τους πολίτες στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Και η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί την, το σεβασμό του, των ευρωπαϊκών νόμων και κανόνων όταν ένας πολίτης μετακινείται από μία χώρα στην άλλη. Αυτό εννοούμε το, την προστασία των δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Άρα λοιπόν Ευρωπαίοι πολίτες δεν είναι μια διαφορετική τάξη, δεν δημιουργούμε μια διαφορετική ομάδα Ευρωπαίων πολιτών, ούτε περιορίζεται ή ε, εφαρμόζεται μόνο στις Βρυξέλλες, η οποία πολλές φορές ονομάζεται η πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ε, μιλάω θεωρητικά για, την, ε, για τις θεσμικές Βρυξέλλες δεν είναι το κέντρο του κόσμου οι Βρυξέλλες, όπως η αρχαία Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη. Απλώς είναι το, η, έδρα, η έδρα όλων των στελεχών που προσπαθούν να βελτιώσουν ε, τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και ε, την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Άρα λοιπόν η ευρωπαϊκή ηθαγένεια δεν είναι κάτι καλύτερο ή κάτι χειρότερο από τις εθνικές ηθαγένειες. Ευχαριστώ για να επανέλθω στις διαδικασίες επί παραβάση. Ελπίζουμε να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ χρήσιμες. Ε, θα επανέλθουμε την επόμενη, θα έρθουμε την επόμενη εβδομάδα από μια ερευνητική επιτροπή στη Γαλλικία για την οποία είχαμε πολλές καταγγελίες περιβαλλοντικής φύσεως. Ένα πράγμα το οποίο μας πάει πίσω πριν από 20 χρόνια. Είχαν γίνει διαδικασίες επί παραβάση τότε από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε οι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ να κινηθούν και να αρχίσουν επιτέλου να έχουν ε, σταθμού επεξεργασία, λιμάτων κλπ αν ε, όλες οι ενώσεις ε, τοπικές, περιφερειακές, ε, ψαράδων για παράδειγμα που δουλεύουν, που αλλιεύουν σε διάφορα μέρη, νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα είχαν πάει τόσο καλά και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο δεν θα είχε υπάρξει πρόοδος. Μπορώ όμως να πω ότι έχει γίνει πολύ πολλή δουλειά ε, σε μικρό χρόνο από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, από τη δυστυχή στιγμή βέβαια που άρχισε η διαδικασία επιπαραβάση. Πάντως αυτό συνέβη. Έχετε το λόγο. Η Επίτροπος, κυρία Ρέντι, είπε ότι οι πολίτες αναμένουν συγκεκριμένα δικαιώματα όσον αφορά τις ε, συναλλαγές τους, εμπορικές συναλλαγές στο διαδίκτυο, φθηνότερη περιαγωγή στα κινητά και άλλα. ή, ε, αλλά, ή λιγότερο, οι λιγότερο πλεονεκτικές περιοχές της Ευρώπης ε, έχουν άλλες επιδιώξεις ε, που πολύ διαφέρουν από αυτά τα δύο που ανέφερα. Παραδείγματο χάρη, ε, στις κοινότητες ε, το Ρωμά παραβιάζονται σε μεγάλο βαθμό τα δικαιώματα, υπάρχει στέρηση, εδρεωμένος ρατσισμός εναντίον τους, δηλαδή κατάχρηση σε μεγάλο βαθμό, ε, κακοποίηση και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, δηλαδή ζητήματα πολύ σοβαρότερα από το ανευθυνότερη κινητή τηλεφωνία. Ευχαριστώ. Ξέρετε ότι το πρόβλημα των Ρωμά συνεχώς ανακύπτει στις συζητήσεις μας, ε, πάρα πολύ συχνά. Υπάρχουν ε, πολλά πράγματα που μπορεί να πει κανείς για το θέμα αυτό, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ακόμη και αν δεν είναι τέλεια η κατάσταση, ε, η δική τους περίπτωση λαμβάνεται πολύ συχνά υπόψη. σε σχέση με αυτό που είπατε. Εγώ είμαι από μια μη κυβερνητική οργάνωση που εκπροσωπεί ακριβώς τους Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπόθηκε ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ε, λόγω των μαζικών ε, απελάσεων που έγιναν από τη Γαλλία ε, μας δείχνει το επίπεδο της διάκρισης εναντίον των πολιτών αυτών το 2012 θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε κατά πόσο τα ευρωπαϊκά όργανα θα σκίσουν πίεση στα εθνικά σώματα ισότητας για να υπάρξει ευαισθητοποίηση τα δικαιώματα των Ρωμά ή αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκοπό να αναλάβει άλλου είδους δράση για να μην ε, την χάνουν διακρίσεων τα δικαιώματα των Ρωμά να δώσω το λόγο ίσως κυρίως στον κύριο, στον κύριο Νεμίτς. Ε, έχετε το λόγο. Yes, thank you very much. Um, ε- Ευχαριστώ. Ε, έχουμε παρουσιάσει μια έκθεση αξιολόγηση σε σχέση με την πρόοδο για τα θέματα Ρωμά στις 21 Μαΐου του 2012. Ε, η έκθεση αυτή έχει όντως δείξει ότι πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα όσον αφορά την εξασφάλιση χρηματοδότησης ε, για την ένταξη των Ρωμά και την ύπαρξη παρακολούθησης των διακρίσεων κατά των Ρωμά. Νομίζω ότι η σαφής απάντηση στην ερώτησή σας είναι ναι. Είμαστε σε διάλογο με τα κράτη-μέλη. Έχουμε δημοσιεύσει την έκθεση αυτή και νομίζω ότι θα ήταν δίκαιο να πει κανείς ότι η ε, τρέχουσα επιτροπή υπό την ηγεσία ε, του Προέδρου της Βαρόσο και της Αντιπροέδρου Ρέντινγκ είναι υπέρ ε, της προάσπισης των δικαιωμάτων και της εξασφάλισης των δικαιωμάτων των Ρωμά στα διάφορα κράτη-μέλη και υπάρχει άλλωστε και ένα σχέδιο δράσης, μια στρατηγική υπέρ των Ρωμά που θεωρήθηκε μάλιστα και η πιο ενεργός που έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια. Κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Not least the one about the right to good administration because... Θα ήθελα να σχολιάσω, λέει η κυρία Λαμπέρτ, για το θέμα της αντιμετώπισης από πλευράς ε, διοικητικών αρχών η, όσον αφορά η έναρξη διαδικασίας ε, προσφυγής για παραβίαση δικαιωμάτων κλπ. Ε, ε, σε περιπτώσεις μεγάλης καθυστέρησης ανταπόκρισης σε διοικητικά αιτήματα και ξέρω ακριβώς τέτοιες περιπτώσεις, αυτές όλες οι διαδικασίες δίνουν ε, καινούργια δικαιώματα στους Ευρωπαίους πολίτες αλλά επίσης ε, έχουμε αποφασίσει ότι θα πρέπει να δίνεται και κατάλληλη εκπαίδευση κατάρτιση στις αρμόδιες αρχές όσον αφορά την αποφυγή διακρίσεων, τη διευθέτηση υποθέσεων κοινωνικής ασφάλειας κλπ. Τώρα για τις συντάξεις βεβαίως υπάρχουν αυτά τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα καθορισμού των συντάξεών τους. Αλλά είναι σαφές ότι σε πολλές περιπτώσεις οι συνταξιούχοι τη χάνουν ε, ε, πάρα πολύ κακής, ε, απέσιασε θα έλεγα μεταχείριση από πλευράς αρχών και πρόσβαση στις συντάξεις τους είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, θέμα προτεραιότητος, διότι πολλοί ε, συνταξιούχοι ε, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στη σύνταξή τους ή δυσκολεύονται ιδιαίτερα επειδή δεν υπάρχουν οι κατάλληλες ε, διασυνοριακές συμφωνίες. Όλα αυτά τα θέματα δείχνουν πόσο σημαντικό είναι το πρόγραμμα προβολής των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών και η Επιτροπή Επασχόληση Κοινωνικών Υποθέσεων φέτος θα αναθεωρήσει όλη το, όλο το πλαίσιο της νομοθεσίας αποφυγής αρνητικών διακρίσεων στον τομέα της εργασίας και επίσης θα εξετάσουμε την πρόσβαση σε περίθαλψη, σε, προ, σε υπηρεσίες υγείας ε, και θα εξετάσουμε επίσης ε, και την κατάσταση στα κράτη-μέλη ότι όπου υπάρχουν κονδύλια τους Ρωμά αλλά όπου γίνεται η επιλογή να μην χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια αυτά. Θα ήθελα, λέει η κυρία Μακδόνελ, να πω και εγώ μετά από όλα αυτά που ελέγχθησαν για τη σχέση μεταξύ των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της χάρτας θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ηθαγένειας. Ε, είναι αλήθεια ότι όλη η συζήτηση που οδήγησε στην σύνταξη της, του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων στόχευε και μέσω του τύπου και των δημοσίων σχέσεων να επιστήσει την προσοχή στους Ευρωπαίους πολίτες στα θέματα αυτά. Τώρα βεβαίως ε, η υλοποίηση είναι δεσμευτική η βάση της συνθήκης της Λισαβάνας και η κατάσταση έχει γίνει πολύ κρίσιμη διότι πολλές προσφυγές γίνονται τώρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε αποφάσεις του είναι εξαιρετικά προσεκτικό στις σχέσεις αυτή που υπάρχουν με, μεταξύ συνθήκης και εισαγένειας Και ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις το δικαστήριο έχει αποφανθεί. Εάν αυτή η περίπτωση είναι εκτός ε, αρμοδιότητος ε, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας τότε θα πρέπει να προσφύγει ο πολίτης ή οποιοδήποτε τέλος πάντων ε, στο βάση του, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, πολύ ισχυρέ διαδικασίες οι οποίες ε, υπάρχουν και σε άλλους οργανισμούς. Ξέρω βεβαίως ότι πολλοί πολίτες επισημούν να, ενδυ... να ενδυναμωθούν ακόμα περαιτέρω οι σχέσεις μεταξύ των δικαιωμάτων των πολιτών και του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και αυτό ίσως θα μπορούσε να το συμπεριλάβει η Κομισιόν στην επόμενη έκθεσή της. Ευχαριστώ πολύ. Νούλα Μόλ λέγομαι. Είμαι νομικός ε, στο Air Center και θα ήθελα να συνεχίσω από κάτι το οποίο αναφέρθηκε ασαφώς ε, με, από κάποιους ομιλητές ε, σήμερα το πρωί. Έχουν περάσει 24 χρόνια από τα συμπεράσματα του Τάμπερε, τα οποία αποφάσισαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες δράσεις, ώστε οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα χαίρουν των ε, ίδιων κανόνων, με στόχο να έχουν ένα καθεστώς το οποίο προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο ε, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και 24 χρόνια αργότερα δεν νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει και πάρα πολύ. Ε, παρά το γεγονός ότι η οδηγία για την επανένωση των οικογενειών και των ε, ε, μακροχρόνια ε, ε νόμιμος δια, κατοίκων που διαμένουν στη χώρα έχουν κάνει κάποια πράγματα, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά δεν επέτρεψε να προχωρήσουν αυτές οι οδηγίες και επέμενε ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλο ποσοστό ε, διακριτικής ευχέρειας στα κράτη-μέλη και δεν θεωρώ ότι έχουν προχωρήσει όσο θα έπρεπε. Οι πολίτες αυτοί οι οποίοι διαμένουν ε, ε, για μεγάλο χρονικό διάστημα στη χώρα πληρώνουν τις ίδιες εισφορές και τους ίδιους φόρους με τους υπόλοιπους ε, κατοίκους της χώρας αλλά δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και θα ήθελα να ξέρω γιατί ακριβώς αναφερόμαστε το 2013 για πολίτες με πι κεφαλαίο που είναι οι πολίτες οι οποίοι απολαμβάνουν τα δικαιώματα του κράτους μέλους και τι γίνεται με τους πολίτες ε, οι οποίοι έχουν ε, τις ίδιες ευθύνες, τις ίδιες ε, οικονομικές δυσχέρειες και τα ίδια, και τα ίδια οικονομικά βάρη, αλλά αποκλείονται από κάποια προνόμια και κάποια ωφέλη. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική ευρωπαϊκή ηθαγένεια και όχι μια ηθαγένεια που αποκλείει κάποιους. Ο κύριος Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι μετά από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, ποικιλόμορφη συζήτηση, θα ήθελα να προσκαστήσουμε να ε, καταρτήσουμε μια χάρτα η οποία θα επικεντρωθεί περισσότερο σε διαφορετική οργάνωση για διάφορα γεωγραφικά επίπεδα. Και υπάρχουν μια σειρά από πράγματα τα οποία ακούστηκαν, τα οποία νομίζω ότι προσανατολίζονται προς ε, αυτή την κατεύθυνση. Λένε ναι, πρέπει να το εξετάσουμε περαιτέρω. Ζητούν ακόμα και νομική απλούστευση, κάτι το οποίο με εκπλήσει, διότι εγώ νόμιζα ότι τους άρεσε αυτό το σύνθετο στοιχείο. Ε, κυρίως ως προς το πώς επικοινωνούμε με τους πολίτες σε ε, τοπικό επίπεδο και η ανάγκη για καλύτερη επικοινωνία. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν υπάρχει ένας κατάλογος δικαιωμάτων που ε, πάνε πέρα της ελεύθερης κυκλοφορίας και το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ηθαγένεια είναι κάτι πολύ παραπάνω από τα δικαιώματα. Ε, είναι αυτή η αίσθηση του ανήκεινο όπως ακούσαμε από τον εκπρόσωπο της γερμανικής ηθαγένειας. Και νομίζω από τη συζήτηση προκύπτει ότι υπάρχουν και τρεις ε, ε, ιδιαίτερα προβληματικοί τομείς στους οποίους θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Καταρχάς ε, το γεγονός ότι υπάρχουν θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά υπάρχουν επίσης και δικαιώματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητα των ανθρώπων, περιβαλλοντική νομοθεσία όπως αναφέρατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, διατάξεις της εσωτερικής αγοράς και πώς συνδέουμε μια πολύ απλή χάρτα και όλο αυτό τον όγκο ε, των στοιχείων που μπορεί να προκύψουν από τους πολίτες και από την νομοθεσία σε όλο το, το φάσμα. Αυτό είναι το ένα μείζον θέμα. Ε, το άλλο ε, μείζον θέμα το οποίο μόλις αναφέρθηκε νομίζω είναι ο κίνδυνος αν πιέσουμε πάρα πολύ την ευρωπαϊκή ηθαγένεια και ενισχύσουμε το χάσμα μεταξύ υπηκών τρίτων χωρών. Και νομίζω ότι τη δώσατε μόνοι σας την απάντηση. Πρέπει να αναβιώσει το Τάμπερε. Έγιναν κάποιες ε, απόπειρες να αναβιώσει το Τάμπερε, αλλά ήταν ε, μεμονωμένες και δεν είχαν καλό αποτέλεσμα. Και από εκεί και πέρα ε, το τρίτο στοιχείο είναι να παραδεχτούμε σαφώς ότι δεν γνωρίζουμε το πεδίο εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή ηθαγένεια αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, έγιναν πάρα πολλές συζητήσει για μειονότητε, για μένα, ε, οι μειονότητε υπάρχουν. Αναφέρονται στο άρθρο 2 της συνθήκης και δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε αυτό. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι ε, ε αυτή τη στιγμή είναι ευρωπαϊκή ηθαγένεια να εξελίξει όλη η διαδικασία. Δεν ξέρουμε μέχρι πού είναι το εύρο τη και θα πρέπει να το δούμε ε, στην πορεία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βενάμπ. Βλέπατε ορισμένα πράγματα εν είδη σύνοψης. Φτάνουμε στο τέλος της ανταλλαγής απόψεων στο πλαίσιο αυτού του πάνελ. Ε, βλέπουμε πόσο ε, δρόμο έχουμε ακόμη για να δώσουμε ψυχή σε αυτή την Ευρώπη ώστε οι ε, Ευρωπαίοι πολίτες να αισθάνονται πραγματικά καλά μέσα σε αυτήν. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που ακούσαμε ε, και θα συνεχίσουμε να τροφοδοτούμε κατά αυτόν τον τρόπο τη σκέψη μας και σε επίπεδο Επιτροπής αλλά και σε επίπεδο Κοινοβουλίου με όλους τους εταίρους μας και τους συνομιλητές μας. Χρειαζόμαστε ίσως πολύ περισσότερη ενημέρωση, πολύ περισσότερη εκπαίδευση, πολύ περισσότερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών ε, και μεταξύ των συνομιλητών μας. Ε, έχουμε στη Γαλλία μια πρωτοβουλία, ε, μια, μια ημερίδα πρωτοβουλίας για τα, τους νέους 16 ετών. Νομίζω ότι ίσως θα έπρεπε να κάνουμε κάτι τέτοιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μπορεί ένας ε, ε, Γάλλος 16χρονος ε, να γνωρίσει άλλους 16χρονους από άλλα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, για τις ομιλίες σας. ένας, ένα από τα δικαιώματα που αποκτήσατε συμμετέχοντας στη σημερινή ακρόαση είναι να φάτε το ελαφρύ γεύμα που βρίσκεται έξω από την αίθουσα, αλλά να διατηρήσετε το μπάτζ σας, ε, πρέπει να τους το δείξετε αν ε, ε, θέλετε να βγείτε από το κτίριο για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να μπορέσετε να ξαναμπείτε μετά, γι' αυτό το λέω. Δυόμιση ώρα θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ. Άρκετ Σιώδη